Πρώτα απ' όλα να δούμε την ημερήσια διάταξη. Θα σα έλεγα να συζητήσουμε το σημείο 8 τη ημερήσιας διάταξη, δηλαδή το στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει τι αναπτυσσόμενε χώρε να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει που συνδέονται με την επισητιστική ασφάλεια, σημείο που προβλεπόταν προ συζήτηση αύριο το πρωί, από το 10 τον αριθμό 10, να το δούμε πριν το 8, γιατί ο κύριος Ταραμπέλα θα πρέπει να μας αφήσει αύριο στις 11.40. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσει, με αυτή τη μόνη αλλαγή στην ημερήσια διάταξη, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα και αύριο. Εάν δεν υπάρχουν παρατηρήσει, τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων θεωρούνται εγκεκριμένα. Να σας πω ότι σήμερα είμαστε και στο διαδίκτυο στη συνεδρίασή μας και υπάρχει και αίθουσα ακρόασης. Η αυριανή συνεδρίαση το απόγευμα θα γίνει στην αίθουσα P1HS001. Θα αλλάξουμε αίθουσα λοιπόν το απόγευμα. Καλώς ήρθατε όλοι. Καλώς ήρθε και ο Επίτροπος, ο κ. Τσόλος. Και να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνεδρία, θυμίζοντας την περασμένη εβδομάδα εκπροσωπήθηκε το Ευρωκοινοβούλιο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας, που πολύ καλά οργάνωσε η Βελγική Προεδρία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επόμενη μεταρρύθμιση τη ε, ΚΑΠ, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του πρώτου πυλώνα και την ευελιξία παρέμβαση λόγω των ε, ιδιαίτερων αναγκών των τοπικών ε, καταστάσεων και των διάφορων δυναμικών. Το Ευρωκοινοβούλιο ήδη έχει τοποθετηθεί για το θέμα αυτό με την έκθεση που εγκρίναμε την έκθεση του κυρίου Λάιεν. Για να εκπροσωπήσουμε το πνεύμα της Επιτροπής μας όμως θέλαμε να μην ε, προκαταβάλουμε το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής και με τον υπολογισμό της δημοσιονομικής κατανομής των κονδυλίων προκειμένου να είναι τα πράγματα μεταξύ των εθνικών αντιπροσωπιών θέλαμε να μπορούμε να αποφασίσουμε τι θα γίνει με την κοινή αγροτική πολιτική στο μέλλον, προκειμένου να είναι ισορρόπη και αποτελεσματική και να ανταποκριθούμε στι μεγάλε παγκόσμιε προκλήσει, στι προσδοκίε των πολιτών και των Ευρωπαίων γεωργών. Είμαι βέβαιο ότι είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε το ρόλο που μα αρμόζει ω συνομοθέτε, αναλαμβάνοντα τι ευθύνε μα στο ευρωπαϊκό πνεύμα και συνεργαζόμενοι σωστά με, με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Περιμένουμε τώρα την επερχόμενη 17η Νοεμβρίου, όπου ο Επίτροπος μας και πάλι στην ε, δική μας Επιτροπή θα παρουσιάσει τη σχετική ανακοίνωση για να ξεκινήσει αυτό το έργο που θα μας απασχολήσει τα επόμενα δύο χρόνια. Πολύ ωραία. Ας αρχίσουμε αμέσω λοιπόν με ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας για το 2011 πρόγραμμα ήδη ιδιαίτερα πλούσιο, από το φθινόπωρο αυτό κιόλα, και με πολύ σημαντικά θέματα τα οποία βρίσκονται επιτάπητος ε, για την ποιότητα, για τα μέτρα του λεγόμενου πακέτου γάλακτος, που ελπίζουμε να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Επίσης θα μας ενημερώσει για το στρατηγικό πλαίσιο που πρόκειται να υιοθετηθεί για καλύτερο συντονισμό μεταξύ της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου και των υπόλοιπων διορθωτικών πολιτικών. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Τσόλος αμέσως για να ξεκινήσει η συζήτηση για ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή. Παρακαλώ. Euh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη κάνατε ένα τμήμα αυτών που ήθελα και εγώ να κάνω παρουσιάσατε κάποιες προτεραιότητες της Επιτροπής από τώρα μέχρι το τέλος του χρόνου. Έτσι βεβαίως δείχνουμε και ότι υπάρχει εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας πω ότι σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά με καλείτε εδώ στην Επιτροπή. Είναι πολύ ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ ημών. Παρ' όλα αυτά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασιών μας. Κάτι που εγγράφεται στα πλαίσια της Λισαβόνας και της παρουσίασης που έκανε ο πρόεδρος Μπαρόζο στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το πλαίσιο αυτής της γεωργικής πολιτικής. Στις 17 Νοεμβρίου θα είμαι εδώ πάλι και θα αναφερθώ στην καυτή ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον της ε, ΚΑΠ. Αυτό θα το κάνω μόλις βγω από την συνεδρίαση της Επιτροπής η οποία θα υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές για να ξεκινήσουμε έναν διάλογο για το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι από τώρα μέχρι το τέλος του 2010 να προχωρήσουμε, να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε προτείνει που έχει συζητηθεί με τις πολιτικές ομάδες της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα βάση της συνθήκης της Λισαβόνας μέχρι το τέλος του 2010. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να υποβάλουμε αυτή την διαδικασία σύμπλευσης με τους τέσσερις πιο σημαντικούς κανονισμούς κοινή οργάνωση των αγορών, ανάπτυξη πέθρου, χρηματοδότηση της ΚΑΠ και άμεσες πληρωμές. Τα πράγματα λοιπόν έχουν ξεκινήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και θα είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τις προτάσεις μας για την ανάπτυξη της υπαίθρου και οι δύο άλλοι κανονισμοί θα ακολουθήσουν όσον αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και την χρηματοδότηση της κοινή αγροτικής πολιτικής. Βεβαίως όσον αφορά όλα τα θέματα αυτά υπάρχει η ρύθμιση της παραγωγής, η φρουτοχημή, καθώς και όλα τα άλλα θέματα που θέλουμε να καλύψουμε Το 2011 θα ακολουθήσουν οι κανονισμοί, ίσως λιγότερο σημαντικοί οι κανονισμοί, οι οποίοι όμως επίσης θα πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της κοινή αγροτικής πολιτικής. Όπως ξέρετε, το νομοθετικό έργο είναι πολύ σημαντικό, αλλά μέχρι το τέλος του 2010 θέλουμε ήδη να σας δώσουμε κάποιες πρώτες προτάσεις έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και η δική σας δράση στην κοινή αγροτική πολιτική. Θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Όπως σας είχα πει και όταν συνάντησα τους υπεύθυνους των πολιτικών ομάδων αυτό το χρονοδιάγραμμα το οποίο καλύπτει το 2010-2011 και εν μέρη το 2012 δεν ακολουθεί αρκούς ρυθμούς. Το έργο που καλούμεθα να επιτελέσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι υπηρεσίες μας λοιπόν εργάζονται από κοινού, προετοιμάζουν την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και το νομοθετικό πακέτο που θα υποβάλουμε το Ιούλιο. Οι ίδιες λοιπόν νομικές υπηρεσίες κάνουν αυτή την εργασία ταυτόχρονα και επαναλαμβάνω από την αρχή του 2011 θέλουμε να υπάρξει αυτή η σύμπλευση για τα πιο σημαντικά στοιχεία της ΚΑΠ. Θα ήθελα να σας διευκρινίσω κάτι που είδαμε στον τύπο όσον αφορά την κοινή επιστολή που έστειλα με τους επιτρόπους Χάντα Μανάκη και Άντοβερ. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα πιλωτικού σχεδιασμού για τα Ταμεία Συνοχής, Κοινωνικό Ταμείο και Αλίας. Και θα ήθελα ευθύς εξ αρχής αν αυτό δεν ήταν σαφές, να σας διαφημίσω ότι δεν πρόκειται για εγκατάληψη του προγράμματος για την ανάπτυξη της υπαίθρου προς όφελος μιας ενιαίας προσπάθειας ενίσχυσης των διαστροτικών ταμείων. Το κάθε ταμείο παραμένει με ξεχωριστούς στόχους, με ξεχωριστή υλοποίηση. Απλώς εμείς προτείνουμε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τον συντονισμό αυτών των τεσσάρων ταμείων. Όταν ήρθα για τις ακροάσεις πριν ε, τον διορισμό μου, το είπα με μεγάλη σαφήνεια κατά την άποψή μου, η ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να βρει τη θέση της και έχει τη θέση της στα πλαίσια της ΚΑΠ. Θέλω όμως καλύτερο συντονισμό με τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία και αυτό εξυπηρετεί την υλοποίηση της κοινή αγροτικής πολιτικής, την υλοποίηση της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου. Στόχος μας είναι να μην υπάρχουν ασαφή σημεία, γκρίζες ζώνες, δηλαδή πολιτικές που δεν καλύπτονται από κανένα ταμείο και να αποφύγουμε και επικαλύψεις που πολλές φορές δημιουργούν, σε κάποιες, δημιουργούν κάποιες παρεξηγήσεις και καταχρήσεις σε τοπικό επίπεδο. Αλλά και για όλους οι οποίοι αποφελούνται είτε πρόκειται για δήμο, για κοινότητα, είτε για ιδιωτικό φορέα, περιφερειακό ή δημοτικό, να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια συντονισμός και η κοινή αγροτική πολιτική να μπορέσει μέσω της πολιτικής της ανάπτυξης της υπαίθρου να διασφαλίσει μια καλύτερη συνεισφορά όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Θα ήθελα αυτό να είναι σαφές για όλους. Αυτή η πρωτοβουλία η κοινή των επιτρόπων δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο την αναλάβαμε. Τώρα, πρόγραμμα εργασιών μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα άλλο νομοθετικό πακέτο, πολύ σημαντικό, το έχουμε παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι το πακέτο για την ποιότητα. Το Δεκέμβριο το πακέτο αυτό για την ποιότητα θα καλύψει κάποια σημεία της έκθεσης ένα πακέτο το οποίο θέλει να διασφαλίσει την καλύτερη προστασία και τον σαφέστερο ορισμό των γεωγραφικών τόπων προέλευσης αλλά και όλων των σημάνσεων που αφορούν την ποιότητα το ίδιο για τα παραδοσιακά είδη και υπάρχουν και κάποια νέα σημεία τα οποία θέλουμε να συμπεριλάβουμε σήμανση για τα τοπικά προϊόντα και ένα σύστημα για την διάθεση στην αγορά προϊόντων από ορεινές περιοχές μεταξύ άλλων και με αυτό το πακέτο για την ποιότητα και κάποιες απαραίτητες προσαρμογές άλλων κανονισμών θα δημιουργήσουμε τη δυνατότητα διασφάλισης κάποιων ενδείξεων για τον χώρο παραγωγής. Αυτό ζητήθηκε πολλές φορές από μέλη του Κοινοβουλίου. Μέχρι το τέλος του χρόνου και εκ το πακέτο για την ποιότητα θα υποβάλουμε και ένα πακέτο νομοθετικό για το γάλα. Και εδώ, βασιζόμενοι στα συμπεράσματα μιας ομάδας ε, υψηλού επίπεδου, ξέρω ότι και εσείς συζητήσατε το θέμα αυτό εδώ και στο Συμβούλιο. Στόχος μας είναι, με αυτό το πακέτο για το γάλα, να είναι να προσφέρουμε στους παραγωγούς αλλά και σε όλου του οικονομικούς φορείς που δρούν στον τομέα του γάλατος εργαλεία και μέσα έτσι ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν για την περίοδο που θα λήξουν οι ποσοστώσεις στον τομέα του γάλακτος. Και επειδή ξέρω ότι αυτή η απόφαση έχει ήδη ληφθεί, ο τομέας του γάλακτος χρειάζεται κάποιες προοπτικές και κάποια σταθερότητα. Η παραγωγή χρειάζονται αυτήν την σταθερότητα και τις προοπτικές για να μπορέσουν να συνεχίσουν οι επενδύσεις και να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Πιστεύουμε τα μέτρα αυτά, ο συνδυασμός αυτών των μέτρων, η δυνατότητα διαπραγματεύσεων, η ενδυνάμωση των επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και η δυνατότητα ανάθεσης, ο διαπαγγελματικός ρόλος περισσότερη διαφάνεια των οργανώσεων, συγγνώμη, η διαφάνεια και η δυνατότητα όλων αυτών των επαγγελματικών κλαδικών οργανώσεων να περάσουν σε διαπραγματεύσεις και όσον αφορά τις εξελίξεις στον τομέα των τιμών και των ποιοτικών προδιαγραφών πολύ συγκεκριμένες προτάσεις θα υποβληθούν. Είχα πει επίσης ότι το Νοέμβριο θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία διαβουλεύσεων. Το Κοινοβούλιο βεβαίως και εδώ παίζει ένα σημαντικό ρόλο για το νομοθετικό πακέτο που θα αρχίσουμε να συζητάμε ήδη από τον Νοέμβριο. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά νομοθετικά ε, σχέδια που έχουμε, αλλά πιστεύω ότι θα επανέλθουμε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ εγώ, Δάτσαν. Έχουμε μια μακροσκελέστατο, ένα μακροσκελέστατο κατάλογο αγορητών. Να ξεκινήσουμε με τους πρόεδρους των ομάδων μας, ο κύριος Δέσου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που μας ενημερώνετε εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας και δέχεστε και να συζητήσετε. Εγώ πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι ο συντονισμός και η σύμπλευση θα πρέπει να γίνει πάντα σε σχέση με τη Λισαβόνα και θεωρώ ότι οι κανονισμοί θα συζητηθούν εδώ και θα μπορέσει να παίξει το ρόλο του Κοινοβουλίου όπως προβλέπει η Λισαβόνα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το πακέτο για, για την ποιότητα και αυτά που είπατε για τον τομέα του γάλακτος. Μπορείτε να μας διασφαλίσετε εδώ ότι θα παραμείνουν τα εργαλεία για την οργάνωση των αγορών και ότι τα εργαλεία αυτά δεν θα έχουν σε σκοπό μόνο καθορισμό τιμών, αλλά ότι σε περίοργο κρίσης θα μπορέσουν να παίξουν τον ρόλο τους, γιατί αυτή είναι τελικά και η ουσία και ο ρόλος αυτών των εργαλείων. Όσον αφορά αυτά που διαβάσαμε στον τύπο με την κοινή επιστολή, εγώ δεν πρόκειται να σας δώσω εδώ απολύτως καμία συμβουλή, αλλά πιστεύω ότι τέτοιου είδους περιπτώσεις μπορούν να εξελιχθούν πολύ πιο ομαλά εάν ε, ε, μια τέτοια επιστολή γίνει γνωστή και εδώ αλλά και σε όλους τους αρμόδιους για τη γεωργία εκ των προτέρων. Αν είχαμε ενημερωθεί νομίζω ότι όλη αυτή η αντίδραση και ο εκνευρισμός θα μπορούσαν να είχαν αποφευκθεί. Και βεβαίως όταν μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα από τον τύπο και με τρόπο ο οποίος δεν είναι σαφής, καταλαβαίνετε ότι ο εκνευρισμό μας είναι πολύ μεγαλύτερος. Χαίρομαι ιδιαίτερα πάντως που μπορέσαμε να σας έχουμε σήμερα εδώ και η πολιτική μου ομάδα αλλά και πιστεύω άλλες πολιτικές ομάδες είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε το διάλογο μαζί σας γιατί πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μπορούν σαφώς να μας οδηγήσουν σε καλή συνεργασία και σε καλύτερες προοπτικές για την κοινή αγροτική πολιτική στην Ευρώπη. Ο κύριος Καπολασάντους. Ευχαριστώ, επιτροπές. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ε, παρουσία σας εδώ. Να σας πω ότι είμαστε προετοιμασμένοι και πρόθυμοι να συνεργαστούμε με την Επιτροπή με τρόπο που θα δείχνει την αφοσίωσή μας για το πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε από την πλευρά της ομάδας των σοσιαλιστών και θέλω να θέσω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα για την επιστολή των τεσσάρων επιτρόπων που μόλις αναφέρατε κι εσείς. Η ομάδα μας προφανώς ικανοποιήθηκε ιδιαίτερα με την επιστολή αυτή. Ήταν μια βασική μας μέρημνα και ήταν στοιχεία που περιλάμβανε, περιλάμβανε και το έγγραφο για τους μελλοντικούς προσανατολισμούς της ΚΑΠ και είχαμε εγκρίνει στην Επιτροπή μας στο παρελθόν, οπότε καλώς και αναφέρθηκαν και γι' αυτό και ικανοποίησαν ιδιαίτερα όλα τα μέλη της ομάδας από ως πρωτοβουλία του Επιτρόπου Γεωργίας. Όμως, πώς πιστεύετε ότι μπορούν να υλοποιηθούν τα απαραίτητα της διάρθρωσης μεταξύ των διαφόρων αυτών νέων μέτρων. Στην πράξη θέλαμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Και ένα ερώτημα περισσότερο πολιτικού χαρακτήρα. Την περασμένη εβδομάδα, με ένα δικαίωμα που είναι τελείως της δικής σας ευχέρεια, δύο υπουργοί δύο των, από δύο τα μεγαλύτερα κράτη της Ένωσης τοποθετήθηκαν σε σχέση με το έγγραφο αυτό, που σε σχέση με το δόγμα που εκφράζει ιδεολογικά βρίσκει σύμφωνο στους σοσιαλιστές σχεδόν πλήρως, όμως δεν μπορούμε και να παραναδιδρούμε στο έγγραφο αυτό, συνεισφέροντα επικοδομητικά. Οι υπουργοί λοιπόν τη Γαλλία και τη Γερμανία είπαν ότι πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, πριν από οποιοδήποτε κριτήριο κατανομή των ε, επιδοτήσεων και πριν γίνει οποιαδήποτε επιλογή, θα πρέπει η ποσοστιαία κατανομή του προπολογισμού να μείνει όπω έχει και στο μέλλον. Αυτό μου φαίνεται τελείω ασυνεπε και πάρα πολύ είναι για όλους όσους ε, θεωρούν ότι η ΚΑΠ στο μέλλον θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη, πιο ε, ισότιμη και πιο σωστά ε, μοιρασμένη μεταξύ των γεωργών των διαφόρων κρατών μελών. Αυτό λοιπόν θα προκαθαρίσει την μελλοντική συζήτηση, πιστεύω. Και τέλος, Επίτροπε, να πω ότι σε σχέση με τις προγραμματισμένες μας δραστηριότητες θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα απρόπτα που μπορεί να συμβούν, τα μη προβλέψιμα γεγονότα. Υπάρχει μια τάση αύξησης των δημητριακών που στη χώρα μου τουλάχιστον ιδίω στην προβολή στον τύπο προς το κοινό έχουν ε, ιδιαίτερη επιτυχία. Αυτό λοιπόν με τις τιμές ε, ελπίζω να το παρακολουθεί η Επιτροπή, τις εξελίξεις στην αγορά δηλαδή. Διότι αν έχουμε μια νέα αυξητική τάση των τιμών, θα πρέπει να προβλέψουμε κάτι για να ανταποκριθούμε. Ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε, Λουίς. Ο κύριος uh, και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο. Το πρόγραμμα που μας παρουσίασε είναι αρκετά φιλόδοξο. Θα ήθελα να επικεντρωθώ καταρχήν σε θέματα χρονοδιαγράμματος. Οι, πράξεις, πράξει εφαρμοστικές πράξεις που θα υποβάλλεται και η ανακοίνωση για την ΚΑΠ πιστεύετε ότι δεν θα ε, τροποποιήσουν το χρονοδιάγραμμα, θα καταφέρετε να το σεβαστείτε, γιατί είναι πολύ σοφόρτος. Ε, ε, οι εφαρμοστικές πράξεις που είναι απαραίτητες λόγω της συνδίκης Λισαβόνας πιστεύετε ότι θα περάσουν γρήγορα και χωρίς προβλήματα από, το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, στρατηγική συμφωνία με τους άλλους επιτρόπους. Μπράβο, πολύ καλή αυτή. Να θεωρήσω ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και την υποστήριξη της πρότασης Κομισιόν για τον προϋπολογισμό στις διάφορες ε, πτυχές της. Μια και πρόκειται για στρατηγική συμφωνία περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό. Τρίτον, ε, το, πακέτο για τις λιγότερο προνομικές περιοχές. Υπάρχει κάποια ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα Έχετε τους χάρτες φαντάζομαι από τα περισσοτερα κρατημέλη. Έχουμε τα καινούργια δύο γεωγραφικά κριτήρια. Δεν ξέρω αν όμως πρέπει να, γίνουν και αν πρέπει να γίνει και άλλη δουλειά ή αν σύντομα θα είναι έτοιμη η πρότασή σας. Grazie George. James Nicholson parola. Ευχαριστούμε κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα επαναλάβω κάποια που έχουν ήδη υποθεί. Ε, βέβαια, ελπίζω ότι θα μας δώσετε και λίγο χρόνο, παρόλο που είναι μακρός και κατάλογος των αγορητών. Κύριε Επίτροπε, ξέρετε ότι η Επιτροπή μας θα εργαστεί σκληρά, όχι μόνο τους ερχόμενους μήνες, αλλά και χρόνια αν χρειαστεί για να σας συνδράμει στο έργο σας. Και Έχω την ισχυρή πεποίθηση ότι τώρα πρέπει να προοδεύσουμε, Επιτροπή, από τη φάση της ακρόασης, τη φάση της δράσης. Διότι το να ακούμε και να κάνουμε υποθέσεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο απασχολεί πολλούς. Διότι το θέμα είναι ποιος ακούει και τι καταλαβαίνει αυτός που ακούει. Τώρα η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Επιτροπή μας είναι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας ε, από την πλευρά της συναπόφασης και να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε το μέλλον της μεταρρύθμισης. Πρέπει η ευθύνη αυτή να αναλυφθεί, διότι είναι μια σοβαρή ευθύνη. Και θα πρέπει να επαναλάβω κάτι που είπε και ο κύριος Ντες. Δεν είναι καλό εμείς ως μέλη της Επιτροπής να βλέπουμε δημοσιεύματα στον τύπο όπου προκαταβάλλεται η δική μας η θέση με, άλλη, με δηλώσεις τρίτων. Όχι, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε διαρκώς για σχεδιαζόμαστε αλλαγές. Για συγκεκριμένα ζητήματα. Εγώ απέχω πολύ το να πιστεύω ότι το να συνδυαστεί η ανάπτυξη της υπαίθρου με την κοινή ελευτική πολιτική δεν θα προσθέσει περισσότερο διοικητικό άχθος, δεν θα δώσει λιγότερους πόρους ε, εκεί που πραγματικά χρειάζονται και τα κονδύλια τελικά δεν θα πηγαίνουν στο σωστό προορισμό. Είμαι πολύ λιγότερο πεπισμένο από εσά, λοιπόν, Επίτροπε, και θα πρέπει να κάνετε πολλά για να με πείσετε. Και επίση, ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σα και απλώ θα θυμίσω αυτό που είπε και ο Λουί για τι ισχυρέ διακυμάνσει των τιμών. Οι τιμέ δεν ανησυχούν μόνο του καταναλωτέ στην Πορτογαλία, αλλά παντού. Οι τιμέ του κρέατο των ε, ζωοτροφών ήδη αυξήθηκαν και στη δική μα χώρα και στη δική μου περιοχή συγκεκριμένα την τελευταία Παρασκευή. Και φαίνεται ότι θα αυξηθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς και άλλο τουλάχιστον 5% μέχρι να βγει το 2010. Τι πιστεύετε λοιπόν θα πρέπει να γίνει στο μέλλον σε σχέση με αυτέ τι ισχυρέ διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά. James Martin. Ευχαριστούμε, James, ο κύριος Γεια, Κύριε Κυρία Επίτροπε, πρόκειται για ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, πολύ εκτεταμένο και είναι πάρα πολύ ε, ενθαρρυντικό το ότι θέτεται εδώ τους στόχους με σαφήνεια Θίξατε κάποια θέματα που όπως και ο συνάδελφος Κάπουλος Σάντος είναι πραγματικά φιλόδοξα. Όσον αφορά τις διαβουλεύσεις, τις δημόσιες διαβουλεύσεις όπως τον Ιούλιο, θέματα που αφορούν ιδιαίτερα και την κοινή γνώμη. Πρόκειται για θέματα που δεν είναι απλώς θέματα που αφορούν τα εισοδήματα των αγροτών, αλλά καλύπτουν και πολλούς άλλους τομείς τομείς που ενδιαφέρουν σήμερα την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη και την κοινή γνώμη. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον το ότι ξεκίνησε αυτή η δημόσια συζήτηση και μπορούμε εδώ να εμπλακούμε και εμείς. Η Ήπεθρος αλλά και το δημοσιονομικό πλαίσιο, κάτι που σαφώς και θα πρέπει να συζητηθεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πολιτική στον τομέα της γεωργίας σήμερα συμπεριλαμβάνει και πολλά άλλα σημαντικά θέματα. Το τελευταίο καιρό υπήρξαν εκθέσεις όπως αυτή του Σοσεμποβέ, η μεταρρύθμιση της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής και εγώ θα ήθελα εδώ να δω πώς θα δεχτείτε και θα συμπεριλάβετε στο πρόγραμμά σας τις δικές μας προτάσεις, συγκεκριμένα για το γάλα είναι ένα θέμα που συζητούμε εδώ και πολύ καιρό με έντονο τρόπο και δεν μας ενδιαφέρει μόνο το πώς θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και τους παραγωγούς, αλλά ο έλεγχος της αγοράς, ο έλεγχος των ποσοτήτων και μέχρι να φτάσουμε στις τελικές προτάσεις θα πρέπει να δούμε, θα εγκαταλείψουμε τελείως ε, τη ρύθμιση και τις ποσοστώσεις ή θα βρούμε μια άλλη λύση για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Νομίζω ότι για πολλούς τα θέματα επίσης της ανάπτυξης της υπαίθρου είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ακόμα πολλά ερωτηματικά παραμένουν και αναρωτιέμαι αν έχουμε μια κοινή κατευθυντήρια γραμμή εδώ όσον αφορά το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής, νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο. Και ενώ οι διακυμάνσεις στην παγκόσμιες αγορές είναι σήμερα δεδομένες, θα πρέπει να δούμε πώς τα επόμενα πέντε χρόνια μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σχετική σταθερότητα. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ ανυπόμονοι και Ελπίζω το Νοέμβριο να έρθετε με πολύ πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ελπίζω λοιπόν μας να είναι επικοδομητική. Μέχρι τώρα δείξατε ότι ξέρετε να μας ακούτε και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Φοντάνα. Κύριε Πίτρο, πρέπει να σας ευχαριστήσω διότι είναι πολύ σημαντικό να είστε εδώ για να μας ακούτε, να ακούσετε όσα έχουμε να σας πούμε. Η έκθεση για την ποιότητα του συναδέλφου κυρίου Σκότα ήταν πραγματικά κάτι που σωστά λάβατε υπόψη και θέλω να ρωτήσω το εξή σε σχέση με το πακέτο περί Να υποθέσουμε ότι θα υπάρξει κάτι εσωτερικός, δηλαδή για εισαγωγέ προϊόντων που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν ενδεχομένω την ίδια ποιότητα με τα δικά μας προϊόντα. Δεν υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός εδώ που δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες για όλους τους Ευρωπαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να αναλάβει δράση σχετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να βελτιώσουμε τα πράγματα όσο γίνεται και μάλιστα πολύ άμεσα. Ευχαριστούμε κύριε Φοντάνα και τώρα οι υπόλοιποι αγορητές μετά τους συντονιστές. 16 έχουν γραφεί στον κατάλογο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ μεγάλες οι διαστάσεις της συζήτησης και να δώσουμε το λόγο και στον Επίτροπο για να απαντά. Φαντάζομαι ότι μπορείτε να ακούτε ορισμένους μαζί, αλλά μετά από ένα σημείο θα πρέπει να απαντάτε κιόλας. κυρία Γέγκλε πρώτη. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Γεωργίας κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τόσο νωρίς θέλετε να έρθετε και να συνομιλήσετε μαζί μας. Όταν μιλάμε για το δεύτερο πυλώνα και όταν αναφέρατε το θέμα της κοινή επιστολής με τους άλλους επιτρόπους Θεωρώ και εγώ ότι αυτή η διασαφήνιση ήταν απαραίτητη. Ήταν απαραίτητη για να ξεπεραστούν διάφορες παρεξηγήσεις. Από την άλλη μεριά πιστεύω και εγώ ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να προχωρήσουμε με πολύ πιο σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και προσανατολισμούς. Όπως και άλλοι συνάδελφοι θα συμφωνήσω και εγώ ότι οι συνομιλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές μεταξύ επιτρόπων να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε για το μέλλον να βρούμε κοινέ λύσεις. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Κάπελος, είναι... Ο συνάδελφος Καπόλα Σάντος είναι σημαντικό να καλύψουμε από όλες τις απόψεις τα θέματα αυτά της ανάπτυξης στην Πέθρου. Ε, όσον αφορά τις διμερείς συμφωνίες, κύριε Πίτροπε, παραδείγματος χάρη είναι αυτή που αφορά την Κορέα ξέρω ότι υπάρχουν εξελίξεις. Εγώ είμαι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας με τον Καναδά. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά έχουν ληφθεί τα θέματα αυτά. Είναι πολύ πιο ψηλά στις προτεραιότητες, στον κατάλογο προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα βιομηχανικά θέματα και άλλα θέματα και όχι τόσο πολύ τα γεωργικά που θα έπρεπε να μας αφορούν. Πώς θέλετε να τοποθετηθείτε στο θέμα αυτό εσείς. Θα απαντήσει σε όλους ο Επιτροπός, όμως να δώσω το λόγο σε μερικούς ακόμη συναδέλφους. Θα απαντήσουμε στο πρώτο γύρο ερωτήσεων. Μετά θα ακούσουμε τις υπόλοιπες και μετά θα ξαναπαρέμβει ο Επιτροπός. Ευχαριστώ πολύ, η ε, κυρία Γκαρσία Πέρεθ. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Δεν θα αναφερθώ σε θέματα τα οποία ήδη έθιξαν άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι για το μέλλον της ΚΑΠ έχουμε ήδη ανταλλάξει απόψεις και θα συνεχίσουμε. Ελπίζω ότι στις 17 Νοεμβρίου θα μπορέσουμε να αναλύσουμε πολύ πιο συγκεκριμένα την πρόταση της Κομισιόν. Θέλω να θίξω μόνο ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφέρθηκα σε αυτό και άλλοι συνάδελφοι βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να μας δώσετε απάντηση. Είναι το θέμα το, της τιμής των σιτηρών και το πώς επηρεάζει την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία. Ήδη άρχισε να θίγει τον τομέα της κτηνοτροφίας, ιδιαίτερα στο τομέα των, της εκτροφής χείρων, η αύξηση της τιμής. Είμαι σίγουρη ότι ο Επίτροπος γνωρίζει πως η αποδοτικότητα της εκτινοτροφίας σχετίζεται άμεσα με το κόστος των ζωοτροφών. Οι ζωοτροφές αντιπροσωπεύουν το 65% του συνολικού κόστους της εκτινοτροφίας κατά μέσο όρο. Συνεπώς ε, είναι σημαντικό να δώσουμε μια απάντηση. Να διατηρούμε επαρκή αποθέματα σιτρών έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την διαθεσιμότητά τους σε στιγμές κρίσης όπως αυτή την οποία ζούμε σήμερα. Άκουσα χθε ότι ανελήφθη μια ε, πρωτοβουλία να βγουν τα σιτηρά από την παρέμβαση να βγουν ποσότητε εισιτηρών από την παρέμβαση. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν αν έχει βάση, αν είναι αλήθεια αυτή η φήμη όχι. Ευχαριστώ. Μάρκ Ταραμπέλα. Ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ. Στι 14 Σεπτεμβρίου υπήρξε μια δήλωση τη Γαλλία και τη Γερμανία για την ε, κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013. Το αδύναμο σημείο αυτής της κοινή θέση κατά την άποψή μου είναι ότι θεωρεί το παγκόσμιο πλαίσιο και τη διακυμάνσεις των τιμών σαν κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Μιλήσαμε για τα δημητριακά, αλλά αυτό ισχύει και για το γάλα και για άλλους τομείς των αγροτικών προϊόντων. Θεωρείτε κι εσείς ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να αλλάξουμε, είτε στις 17 Νοεμβρίου θα μας δώσετε κάποιες απαντήσεις για το πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, εξαιρετικά σημαντικές διακυμάνσεις ε, τιμών. Και ελπίζω εδώ στο Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να είμαστε τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμά ε, σύμφωνοι για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο πλήττει σήμερα τους περισσότερους τομείς. Ο Επίτροπος είπε ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να περιορίσουν ή και να ε, απαγορεύσουν τα γενετικά τροπημένα τρόφιμα και τις ε, ζωοτροφές στην επικράτειά τους ε, ακόμα και αν έχει αποφασιστεί ελεύθερη κυκλοφορία τους σε ευρωπαϊκό πεδίο. Οπότε η ερώτησή μου είναι η Κομισιόν δέχεται τις, διαφορέ τις διαφορές στην ανταγωνιστικότητα που θα προκύψουν από αυτό διότι ορισμένα κράτη-μέλη μπορεί να απαγορεύσουν τι γενετικά τροπημένε ουσίε, ενώ άλλε όχι. Αυτό θα δημιουργήσει μια διαφορά, ένα χάσμα σε, στην ανταγωνιστικότητα ο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάποιες χώρες, μειονέκτημα για κάποιες άλλες. Επίσης, πώς βλέπει τη σχέση της Ευρωπαϊκής με το, Διεθνή, Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Τροφίμων, ο Επίτροπος. Ο κύριος Γιάρ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις προς τον Επίτροπο όσον αφορά τον κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Θέλω να κάνω μια έκκληση προς την Επιτροπή, προς τον Επίτροπο. Μιλήσατε για συντονισμό. Αυτό επουδενή λόγο δεν θα πρέπει να σημάνει και επιδότηση της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Πιστεύω ότι θα πρέπει πραγματικά να δώσουμε έμφαση στην ανάπτυξη της υπαίθρου και για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές ιδιαίτερα. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ίσως θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τελείως ξεχωριστά αυτά τα δύο θέματα έτσι ώστε να του δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ο κύριος Νταντέν, ευχαριστούμε Επίτροπο που είστε και πάλι μαζί μας. Εξ ονόματος της ομάδας μου να διαβεβαιώσω τον κύριο Καπούλα Σάντος ότι το έγγραφο των δύο κυβερνήσεων και η στάση μας δεν σημαίνει ότι θέλουμε πίσω τα λεφτά μας. Δεν ζητούμε αυτό. Ζητούμε απλώς διαιτησίες να μην ολοκληρωθούν μέχρι να αποδοθούν τα σωστά χαρτοφυλάκια. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα λοιπόν. Τώρα για το σημείο που έθιξε και ο επίτροπο, ιδίως για το πακέτο του γάλακτος που θα έρθει τώρα το φθινόπωρο, να τονίσουμε τον κατεπήγοντα χαρακτήρα του πακέτου αυτών μέτρων για την Ήπεθρο. Την περασμένη μόλις εβδομάδα έλαβα μια επιστολή που πραγματικά με συγκίνησε από έναν συνάδελφο που ασχολείται με την πρόθεση προϊόντων και έχει εγκατασταθεί στην Ορμανδία και τον ξέρω από όταν ήμασταν φοιτητέ. Έχει πάρει λοιπόν κοινωνική βοήθεια γιατί στην η παραγωγική του εγκατάσταση δεν μπορεί να παράγει αρκετά ώστε να βγάλει τα απαραίτητα για να θρέψει τα παιδιά του. Είναι μια πραγματικότητα λοιπόν αυτή, η οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ακόμη και αν δεν τη συζητάμε ιδιαίτερα στι περιοχέ όπου υπάρχει παραγωγή γάλακτο. Κύριε Επίτροπε, είμαστε δίπλα σα στι προτάσει που κάνετε και έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο κοντά σα αρκεί κάποιοι συνάδελφοι να συνδυαστούν μαζί μας και να μας διευκολύνουν τη ζωή. Διότι άκουσα πρόσφατα ότι για το κρέας από την ε, Αργεντινή ε, οι εκπρόσωποι της ε, Μερκοσούρ καταγράφουν μια πρόταση ε, από τους Ευρωπαίους εταίρους για 400 επιπλέον τόνους που θα έρθουν χιλιάδες τόνους που θα έρθουν προς την Ευρώπη. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν για το εμπόριο κύριε Επίτροπε μας καταστρέφουν την αξιοπιστία. Είναι σαν πισόπλατες μαθηριές. Δηλαδή όλη μας η κοινή αγροτική πολιτική αλλοιώνεται. Ούτε η μεν ούτε η δε δεν θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε με του εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου γιατί θα έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη του. Πρέπει το μήνυμα λοιπόν αυτό να το αντιληφθεί το σύνολο των επιτρόπων, ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι εδώ εκφράζομαι εξ ονόματο όλων των συναδέλφων που είναι μέλη τη Επιτροπή Γεωργία. διότι πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό του απασχολεί και κυρίω μα απασχολεί να προδοθούμε από την ίδια την Επιτροπή. Ευχαριστούμε, Μισελ. Κυρία Ντελάγκερ. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you, Commissioner. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που είσαστε εδώ μαζί μας. Και η δική μου ερώτηση είναι οριζόντια, έχει σχέση με τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά πιο συγκεκριμένα στην πολιτική ανταγωνισμού. Πολλές από τις προτάσεις που κάνετε συνδέονται με την ε, πολιτική ανταγωνισμού, για παράδειγμα, προτάση για το γάλα. Στην έκθεση Μποβέ πολλά από αυτά που ζητούμε δεν μπορούν να θεωρηθούν ως αποκλειστικής γεωργικής αρμοδιότητας. Οπότε, εν ώψη της συζήτησης για την ΚΑΠ, θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποιο μήνυμα από την Κομισιόν ή μια ανακοίνωσή της για το πώς αυτή η συζήτηση για την ΚΑΠ θα συνδυαστεί με μια ευρύτερη συζήτηση για την πολιτική ανταγωνισμού. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σοβαρά την ΚΑΠ χωρίς να συζητήσουμε ταυτόχρονα για την ευρωπαϊκή πολιτική ανταγωνισμού. Και προς το παρόν παίρνω ανάμεικτα σημάδια από την Κομισιόν για αυτό το θέμα. Μήπω θα μα διευκρινιστεί το θέμα αυτό πλευρά Κομισιόν, μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ντελάνγκε. Κυρία Χάνης Γερσία. Ε, Ευχαριστούμε για την παρουσία σας, Επίτροπε. Θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για, το... για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής των ε, ενισχύσεων, παρόλο που δεν μπορείτε να μας δώσετε τα νούμερα. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να μας δώσετε τα νούμερα, μήπως θα μπορούσατε να μας μιλήσετε λίγο για τα κριτήρια τα οποία συζητούν στην Κομισιόν για την αναδιανομή. Ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά την ε, ενίσχυση αναεκμετάλλευση, την επίμαχη αυτή. Ε, θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με την κτηνοτροφία σε χώρες όπως η Ισπανία όπου υπάρχει πολλή κτηνοτροφία χωρίς όμως ε, να υποστηρίζεται από ανάλογη κατοχή γης. Ε, θα, πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης θα ήθελα να γίνει σεβαστή η ε, διαφορά ανάμεσα στις διογραφικές ενδείξεις και στις ενδείξεις προέλευσης. Θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό θα γίνει. Τέλος, ε, τα, ε, θα εξασφαλιστεί ότι τα ποιοτικά αγαθά ε, θα φτάνουν στον καταναλωτή με τους ίδιους όρους είτε είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή από πότε και μετά θα, αρχίσει, θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια ποιότητας και για τα εισαγόμενα προϊόντα ε, Γαβριέλ Ματώ δεν, ο Γαβριέλ Ματώ δεν ε, κατάφερε να γυρίσει από τη Βενεζουέλα ε, γιατί αφαιρέθηκαν τα διαβατήρια ε, από, τις, από του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθυστέρησε λοιπόν και δεν κατάφερε να πάρει το αεροπλάνο. Οπότε ήθελε να, ήθελα να ρωτήσω το εξή. Τι γίνεται με τα προγράμματα ΠΟΣΕΙ και τη συνέχεια του. Είναι πολύ σημαντικά για περιοχέ όπω οι Κανάριε νήσι. Θα μπορούσατε να μα ε, πείτε ποιο είναι το μέλλον του. Ευχαριστώ. Ο Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο που είναι σήμερα εδώ και μπορούμε να έχουμε αυτή τη συνάντηση μαζί του και να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Και εγώ θα κάνω την ίδια ερώτηση όπως και ο συνάδελφος για τις ε, λιγότερο ευνοημένες ε, περιοχές. Εμείς περιμένουμε από την Επιτροπή μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση εκτός της ε, κοινή αγροτική πολιτική και της μεταρρύθμισης. Ένα ξεχωριστό πακέτο. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό γιατί στις λιγότερο ευνοημένε περιοχές υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα, θέματα που σαφώς ε, αφορούν και την επικουρικότητα, και την ευελιξία που έχουν και πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν τα κράτη-μέλη. Γιατί το πιο άκαμπτο σύστημα της, του πρώτου πυλώνα δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες. Και άλλοι δύο συνάδελφοι έθεσαν ε, το θέμα των διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες. Αναφέρθηκε το παράδειγμα του Καναδά. Εγώ θα μιλήσω για το Μαρόκο ακούμε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο προχωρούν. Το Μαρόκο είναι μια πολύ σημαντική χώρα για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οποροκυπευτικά, σημαντικά για τη χώρα μου. Όπως ξέρετε το Μαρόκο χτυπάει και την πόρτα για περισσότερες εμπορικές συναλλαγές Ας μην ανοίγουμε λοιπόν εδώ το παραθυράκι αυτό για μια αγορά η οποία ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες, ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση και τα λαχανικά και τα φρούτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρκετές δυσκολίες έτσι ώστε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τα προϊόντα που έρχονται από άλλες χώρες. Grazie. Ευχαριστούμε. Πραγματικά αυτό το θέμα του Μαρόκου μας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως και μας απασχολεί ακόμη κύριε Επίτροπε. Κυρία Μαγκίνας, το μικροφόνο. Τώρα δουλεύει, αλλά σας ευχαριστώ. Να επαναλάβω λοιπόν τι ευχαριστίες μου προς τον Επίτροπο. Τώρα για τον πολιτικό συντονισμό μεταξύ των Επιτρόπων. Προφανώ θα συμφωνήσω για τα τη εμπορική και γεωργική πολιτική, διότι μεταρρύθμιση τη γεωργική πολιτική δεν μπορεί να μην λαμβάνει υπόψη αυτά που συμβαίνουν παράλληλα στην εμπορική πολιτική και στι διαπραγματεύσει μα. Γίνονται και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίε πολλέ φορέ τρέφονται κατά των Ευρωπαίων παραγωγών και των ίδιων των καταναλωτών. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τα συμφέροντα και των Ευρωπαίων παραγωγών στι εμπορικέ διαπραγματεύσει τι ίδιε. Έπειτα, για το θέμα τη ανακοίνωση που περιμένουμε στις 17 Νοεμβρίου, νομίζω ότι και πάλι αργά είναι η ημερομηνία αυτή. Ήδη μας ανησυχούν κάποια από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την Επιτροπή για τις ενδεχόμενε επιλογές σε σχέση με την κατανομή των πληρωμών. Οι Γεωργοί ήδη ε, έχουν ε, κάποιες υποψίες για το τι θα συμβεί. Ε, ήδη λοιπόν θέλουμε να μας πείτε πόσο μπορείτε να αποσαφηνίσετε τα πράγματα. Είναι πολύ αβέβαιη η κατάσταση. Είναι, υπάρχει κλίμα βεβαιότητας και ανησυχίας και οι γεωργοί προσπαθούν να μαντέψουν τι θα συμβεί. Ε, κάποιοι αισθάνονται ότι έχουν λάβει δυσίωνα μηνύματα. Τώρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ξέρω ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα κρατός μέλος που θέλει να μεταφέρει κονδύλια από τον τομέα αυτό ακριβώς σε άλλους τομείς, γιατί υπάρχουν προβλήματα με τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων αναπτύξης της υπαίθρου. Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά αυτό, σε αυτό το είδους προγράμματα, ή θα μπορεί να συμβεί κατά εξαίρεση για επιμέρους κράτη-μέλη, κάποιοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερα αναπτυξιακά κονδύλια για άλλους τομείς, όπου μπορεί να πάσει και η εθνική τους οικονομία και για τις συμβάσεις ε, που προτείνονται από την ομάδα υψηλού επίπεδου ε, για τις συμβάσεις που απασχολούν κάποια κράτη-μέλη και κάποιους γεωργούς. Μπορεί να αντικατασταθούν πλέον ποσοστώσει από συμβάσεις. Και επίσης, σε σχέση με τη μεταφορά των ζώων θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία του χρόνου, εξ όσων γνωρίζω. Αντί λοιπόν να προβλέψουμε περισσότερη νομοθεσία για τις μεταφορές των ζώων, δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τους υπάρχοντες κανόνες. Η ενίσχυση αυτή πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πριν ε, κάνουμε περισσότερα, διότι κάποιε φορέ το να προβλέπουμε περισσότερα μέτρα επιβαρύνει περισσότερο τα πράγματα αντί να τα διευκολύνει. Θα περιμένουμε πάντω σε κάθε περίπτωση τι αντιδράσει σα και την Παρασκευή Επίτροπε. Ευχαριστούμε ο κύριο Μποβέ. Oui, monsieur le commissaire. Euh, Κύριε Επίτροπε, με συγχωρείτε που άρχισα να φτάσω. Ε, προβλήματα με τα τρένα. Είναι και μια είδηση αυτό όταν τα τρένα καθυστερούν αποτελεί είδηση αυτό και σα φέρνω και την πληροφορία μαζί. Τρία σημεία λοιπόν, το πρώτο ήδη έχει σχολιαστεί. Η έκθεση που επέβαλα προς το Κοινοβούλιο και που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία περιείχε δύο σημαντικότατα, τρία σημαντικότατα σημεία. Πρώτα απ' όλα λαμβάνεται υπόψη το κόστος παραγωγής, έπειτα η ανάγκη διαφάνειας για τους ελέγχους από την επεξεργασία μέχρι τους φορείς μεγάλης διανομής που κατέχουν το περιθώριο της αγοράς αυτή τη στιγμή και έπειτα η καταπολέμηση της κερδοσκοπίας. Πολλοί είναι οι συνάδελφοι που πήραν το λόγο ε, και για το θέμα της ποιότητας. Εγώ θα έλεγα ότι πιο πολύ πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κερδοσκοπία, διότι είναι ξένοι οι που δρούν αυτή τη στιγμή στην αγορά μας και ε, φροντίζουν να κερδίσουν από την αγορά των δημητριακών λόγου χάρη και με συνελλαγέ που μόλι σήμερα μπορεί να έγιναν. 7% των συναλλαγών παγκοσμίω ανταποκρίνονται στι πραγματικέ ποσότητε που διακινούνται στην αγορά. 80, 93% είναι εκτό παραγωγή. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα κονδυλίων εδώ. Και ξέρω ότι και συναντήσατε και το συζητήσατε το θέμα αυτό με τον Επίτροπο Μπαρνιέ και είναι ένα ζήτημα πρωταρχικό κατά τη δική μου άποψη. Έρχεται πριν από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Έπειτα, για το σκέλος της ποιότητας. Ξέρω ότι προσέχετε πάρα πολύ ό,τι αφορά την ποιότητα. Το πρόβλημά μου σήμερα όμως είναι ότι υπάρχει μια σειρά από προγράμματα που καταρτίζονται και σχεδιάζονται στην Ευρώπη και αντίκυνται στην έννοια της ποιότητας ή μπορεί να καταστρέψουν πολλές αγροτικές περιοχές. Συγκεκριμένα σκέφτομαι ένα σχέδιο για σφαγείο που μόλις επισκέφθηκα κιόλα στην κάτω Σαξονία όπου υπάρχει ένα σχέδιο για σφαγείο με πρόγραμμα να σκοτώνονται 27.000 κοτόπουλα, να θανατώνονται 27.000 κοτόπουλα την ώρα. Μιλάμε για κάτι κολοσιαίων διαστάσεων. Σημαίνει ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον ε, 500 έτσι, τέλος πάντων εκτροφία πουλερικών που θα πρέπει να τροφοδοτούν το σφαγείο αυτό. Αυτά λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουν ότι υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις. Πρέπει να προσέχουμε για τέτοιου είδους προγράμματα και από την άποψη την οικονομική και την κοινωνική και την περιβαλλοντική και για την ευημερία των ζώων. Τι είδου γεωργία θέλουμε να δημιουργήσουμε. Και το λέω αυτό χωρίς να σχολιάσω άλλα προγράμματα όπως λόγω χάρη τη Πολωνία, με την εταιρεία Smithfield όπου δημιουργούνται τεράστια εκτροφία χείρων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές βεβαίως αλλά άλλων διαστάσεων. Να προσέχουμε λοιπόν και για τα γαλακτοκομικά χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις, στις διεπαγγελματικές όπως λέτε εσείς. Για να είναι σαφή και διαφανείς θα πρέπει το σύνολο των συμμετεχόντων να εκπροσωπούν πράγματι όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν κάποιες ε, χώρες όπως η δική μου που κάποια επαγγέλματα έχουν ιδιωτικό καθεστώ. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπροσωπούνται άξια όλα τα επαγγέλματα. Για το θέμα των γενετικώ τροποποιημένων οργανισμών που ανακούστηκε προηγουμένω, η πλειοψηφία των 27 κρατών στην συνάντηση τη περασμένη εβδομάδα είπε ότι δεν ήταν υπέρ, για να μην πω ότι ήταν εχθρική προς την πρόταση της του κυρίου Νταλή. Σήμερα αυτό που νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό από το να προωθηθεί η πρόταση αυτή είναι να, να φτάσει η συζήτηση του γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να δούμε κατά πόσο είναι εφικτή η συνύπαρξη. Αλλά να χρησιμοποιήσουμε και τα πορίσματα της εμπειρογνωμοσύνης. Διότι βλέπουμε σήμερα ότι η εμπειρογνωμοσύνη για τους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς είναι ένας τομέας ιδιαίτερα ομιχλώδης και εκεί επικρατούν οι πολυεθνικές. Θέλω λοιπόν να αναλάβει δράση και για αυτό το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όλα αυτά αφορούν άμεσα την αξιοπιστία της ΚΑΠ. Eh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ανιώ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είμαι ήδη στο 11. Η Επιτροπή όμως δεν θα είναι αύριο μαζί μας η μελλοντική νομοθεσία. Κάτι το οποίο σαφώς ε, και μπορεί να μας οδηγήσει σε, περισσότερη, σε ένα καλύτερο κλίμα, ένα κλίμα εμπιστοσύνης, είναι κάτι που σαφώς και θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2012. Ξέρουμε ότι η κατανομή δεν θα έχει γίνει ορθά ούτε τον Ιανουάριο του 2012 και ξέρουμε ότι μέχρι τώρα η αλλαγή για το όλο σύστημα για τα πουλερικά θα στοιχήσει 13 ευρώ για κάθε πουλί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η σημερινή κατάσταση πλήττει αυτούς που εφαρμόζουν την νομοθεσία. Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Ο και μετά ο κ. Κύριε Επίτροπε, παρουσιάζοντας το νέο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, θα πρέπει να βασιστούμε στο κεκτημένο της ΚΑΠ να σα επιστήσω την προσοχή σε ορισμένους τομείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω χάρη στην διαφοροποίηση της ευρωπαϊκής γεωργίας ανάλογα με τις κλιματικές διαφορές, τις δομικές διαφορετικές διαφορές. Δεν θα μπορούσαμε να ομοιογενοποιήσουμε την κοινή αγροτική πολιτική κατά τρόπον ώστε να μην πληγεί η αποτελεσματικότητά της να έχουμε τα ίδια εργαλεία παρά τις διαφορετικές συνθήκες για διαφορετικά αγροκτήματα και εκμετάλλευσεις. Ένα άλλο ζήτημα, η διατήρηση της γεωργίας και της παραγωγής υπό δυσχερείς συνθήκες. Και δεν μιλώ εδώ για τις ιδιαίτερα ευάλωτες περιοχές, αλλά και για αυτέ όπου υποβαθμίζεται διαρκώ η παραγωγή και τίνει προ εξαφάνιση. Αυτό το είδο η παραγωγή δεν πρέπει να προστατευτεί πριν εξελιχθεί πλήρω. Και κάτι ακόμη που με απασχολεί. Θα δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τα ευαίσθητα θέματα και να μην λάβουμε κανένα μέτρο, διότι στην γεωργία και την κτηνοτροφία υπάρχουν ε, τέτοιες διαφορές, όπως οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματικές διαφορές. Εκεί, αποφεύγοντας την βοήθεια και τη στήριξη, μπορεί να καταστρέψουμε πλήρως μια ολόκληρη αγορά. Οπότε, σε κάποιο βαθμό, περιορισμένο έστω, σαφώς και πρέπει να υπάρχει παρέμβαση λόγω χάρη στην αγορά των δημητριακών. Καμιά σταθερότητα δεν θα καταφέρουμε να έχουμε αν δεν παρέμβουμε. Και ένα άλλο πρόβλημα. Η διέρεση μεταξύ περιφερειακής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Πού αρχίζει το ένα και πού τελειώνει το άλλο. τούμπαλιν. Εάν μιλάμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου, είναι πολλά τα στοιχεία που θα μπορούσαν να μεταφερθούν από αυτή την πολιτική στην ε, περιφερειακή. Σας συγχαίρω μάλιστα και σας ζητώ να μας εξηγήσετε ακριβώς τις ιδιαιτερότητες της κοινή αγροτικής πολιτικής και του κεκτημένου της και σε εμά τους ίδιους τους πολιτικούς όσο και στο κοινό. Διότι κάποιες φορές υπάρχουν ε, άνθρωποι που νομίζουν ότι το γάλα μπορεί να έρθει απευθείας στο κατάστημα χωρίς να έχει βγει από την Αγελάδα. Ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να κάνω πολύ συγκεκριμένη ερώτηση γιατί ο χρόνος πιέζει τον Επίτροπο. Όσον αφορά την έκθεση Σκόδα, η οποία ήταν εξαιρετική το θέμα της ε, σήμανσης και της προέλευσης των προϊόντων. Θα πρέπει σαφώς να ληφθούν μέτρα, ώστε η ποιότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων να είναι εμφανής και να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους καταναλωτές. Το θέμα της μεταφοράς των ζών των ζών. Επίσης ξέρω ότι υπάρχουν πολλά που έχουν γίνει. Το θέμα δεν είναι τα πρότυπα που έχουμε υιοθετήσει. Το θέμα είναι το κατά πόσον αυτά εφαρμόζονται, υλοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές το θέμα είναι περίπλοκο. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητούμε, αλλά καλό θα ήταν η Επιτροπή να μας δώσει κάποια στοιχεία για το προς τα πού οδεύουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Επιτροπέ, για την παρουσίαση των νομοθετικών σας σχεδίων. Να σας ρωτήσω απλώς τα εξής δύο ερωτήματα. Ενώ υπάρχουν πολλαπλές αποδείξεις από τους παραγωγούς βοήου κρέατος και κρέατος αγοπροβάτων, ιδίως το πώς σημαδεύουν τα ζώα αυτά, Υπάρχουν λοιπόν πολλέ ανησυχίε, γιατί εμένα με πλησίασαν Γερμανοί, Βέλγοι και Ολλανδοί κτηνοτρόφοι και μου παρουσίασαν ε, τον ε, διοικητικό γραφειοκρατικό του αγώνα κατά του συστήματο. Ένα έφτασε να μου πει ότι γύρισε πίσω με το κοπάδι του Και ενώ τα ζώα καταφέρνουν να κοιμηθούν, ο εκτροφέας, δηλαδή ο ίδιος, κάθεται επί ώρες μπροστά στον υπολογιστή για να καταφέρει να καταγράψει όσα έγιναν την τελευταία μόλις μέρα. Λένε λοιπόν οι εκτροφείς, οι κτηνοτρόφοι, ότι το σύστημα δεν είναι καθόλου λογικό. Διότι τα δεδομένα ούτως ή άλλως δεν είναι πλήρη <clears throat> και δεν μπορεί κανείς να δει τι έχει γίνει ζώο προς ζώο προηγουμένως. Είναι λοιπόν πολύ ισχυρά αυτά τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει μέτρα για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Ένα άλλο ζήτημα αφορά τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Να ρωτήσω ποια είναι η δική σας άποψη για το ζήτημα αυτό. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι υπέρ της βιοπικιλότητας. Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί ακριβώς αντίκενται σε αυτή την έννοια. Θέλουμε λοιπόν να αποκλειστούν οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί από την λήψη οικονομικής στήριξης. Και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Μποβέ που σχολίασε το θέμα των τεράστιων εκμεταλλεύσεων, των υπέρογκων μεταλλεύσεων. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι η γεωργία γίνεται ένας μεγάλος βιομηχανικός τομέας και αυτό είναι ενάντιο και στην ίδια την ευημερία των ζώων και την ε, υγεία των ανθρώπων φυσικά. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τις ανησυχίες του κυρίου Μποβέ σε σχέση με το θέμα. Mulțumesc. Domnule comisar, trei întrebări scurte și foarte precise. Ați prezentat deja calendarul. Să se facă παρουσιάσατε το χρονοδιάγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις νομοθετικές προτάσεις και ξέρω ότι έγινε και μια πολύ σημαντική συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Νέων Αγροτών που έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προτάσεις σας καθώς η Επιτροπή έχει δείξει ότι θέλει να επανεξετάσει το θέμα της εγκατάστασης των νέων αγροτών. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους νέους αγρότες με πιο αποτελεσματικό τρόπο και θα ήθελα να ξέρω αν προτίθεστε να υιοθετήσετε νέα μέτρα για την στήριξή του. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτή την κοινή θέση της Γαλλίας και της Γερμανίας όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική η Γαλλία και η Γερμανία έχουν μια πολύ συγκεκριμένη θέση όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές που θα πρέπει να καθορίζονται με έναν τρόπο που να έχει σχέση με τους προϋπολογισμούς των κρατών. Δεν μπορώ να κατανοήσω την ε, πρόταση αυτή της γαλλογερμανικής πρότασης. Ευχαριστούμε. Δύο τελευταίες παρεμβάσεις τώρα, κύριο Ζούμπικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπουμε εδώ στην Επιτροπή μας και μάλιστα αρκετά συχνά. Και χαίρομαι που δεν ακούτε μόνο τη φωνή των κυβερνήσεων αλλά και την φωνή των εκπροσώπων του λαού των Ευρωβουλευτών. Εκπροσωπώ τη Λετωνία και ο αγροτικός κόσμος της Λετωνίας ανησυχεί ιδιαίτερα από το γεγονό ότι γίνεται πολλής λόγος για τις άμεσες πληρωμές. Δεν είναι δυνατόν σε κάποιες χώρες αυτές οι ε, πληρωμές είναι 4 έως 6 φορές μικρότερες από τις άλλες χώρες. Υπάρχει μια στρέβλωση λοιπόν και γίνεται λόγος για πλήρη κατάργηση των άμεσων πληρωμών. Κάποιοι λένε από την άλλη μεριά ότι αυτές οι πληρωμές θα πρέπει να συνδέονται με την παραγωγή ενώ κάποιοι άλλοι να μην συνδέονται με την παραγωγή. Θα ήθελα να ακούσω από εσά, κύριε Επιτροπέ. Πώς θα εξασφαλίσουμε μια δικαιοσύνη στον τομέα αυτό. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι γεωργοί της δικής μου της περιοχής ανησυχούν ιδιαίτερα. Και το ίδιο και εγώ. Οι ενώσεις των παραγωγών δεν ενισχύονται αρκετά μόνο διεπαγγελματικά. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές ανισότητες, κέρδη για τις πολυεθνικές και για τις οργανώσεις παραγωγών βεβαίως δεν, με τις οργανώσεις παραγωγών δεν επέρχεται ισορροπία, πλήττονται μικρή παραγωγή. Και βεβαίω υπάρχει και η τάση εξισορρόπηση τη αγορά με τον έλεγχο τη προσφορά. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσετε τη δήλωση του Επιτρόπου που λέει ότι πρέπει να αποδεχτούμε ότι θα έχει λιγότερα κονδύλια η ΚΑΠ. Στην πρόσφατη ακρόασή του στην ε, Επιτροπή για τις Περιφέρειες το είπε αυτό. Έπειτα, πιστεύετε ότι τα μέτρα ρύθμισης της αγοράς πού θα φτάσουν οι συμβάσεις πώς ε, θα επηρεάσουν τις σχέσεις γεωργών και όσων εργάζονται στην βιομηχανία επεξεργασία των ε, προϊόντων. Αυτό πώς το εξετάσει η ομάδα E κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τι άμεσε πληρωμέ στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όπω όλοι γνωρίζουμε, και είμαι σίγουρο ότι το γνωρίζετε κι εσεί, κύριε Επίτροπε, οι άμεσε πληρωμέ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας μόνο εν μέρη φτάνουν στους γεωργούς. Και μάλιστα αυτή η κατάσταση θα παραμείνει όσο έχει μέχρι το 2016 από ό,τι φαίνεται, από ό,τι έχει προβλεφθεί. Το θέμα αυτό έχει θυγεί επανειλημμένο στο παρελθόν στην Επιτροπή μας και είχα την εντύπωση ότι οι συνάλφοι διαφωνούν με αυτή τη διάκριση αυτή τη διακριτική μεταχείριση. Η Κομισιόν σκοπεύει να καταργήσει αυτή την πρακτική. Σκοπεύει η Κομισιόν να φτάσει στο μέγιστο των πληρωμών για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Γιατί οι Γεωργοί είναι από τους πιο φτωχούς ανθρώπους της χώρας μας. Μόρβε, αλλά παρόλα, πρέγω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σε ό,τι αφορά την Ουγγρική Προεδρία το 2011, ποιες είναι οι προσδοκίες σας, οι βασικές σας προσδοκίες και ως Επίτροπος Γεωργίας, σε ποιους τομείς περιμένετε να χρειαστεί περισσότερη συνεργασία από πλευρά Ουγγρική κυβέρνηση και Ουγγρών ηθινόντων, των υπευθύνων δηλαδή για την αγροτική πολιτική. Όσο για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. σε τι φάση πιστεύετε ότι θα έχουμε φτάσει στο εξάμεινο τη Ουγγρική Προεδρία και ποια θα είναι τα βασικότερα ζητήματα, οι βασικέ προτεραιότητε. Οι Ούγγροι Γεωργοί, οι οικογένειε του, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει περιμένουν πολλά από αυτή τη μεταρρύθμιση. Θέλουν να είναι ενεργοί συμμετέχοντε στην αγροτική πολιτική τη Ευρώπη. Γι' αυτό θέλω να ρωτήσω και το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στα λόγια και στι ομιλίε που εκφωνούνται, ε, τονίζει την ανάγκη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ε, με του δημόσιου φορεί στην ε, διαδικασία λήψη αποφάσεων. Πώ να προετοιμάσουμε εμεί του Ούγγρου πολίτε για την Ουγγρική Προεδρία, ξέροντα ότι βεβαίω αυτό είναι και ευθύνη κυβερνητική, αλλά ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλει να συνεργαστεί με του Ούγγρου γεωργού, θα πρέπει να έχει προλύνει το έδαφο. Τελευταία ερώτηση τώρα. Για την ε, διάκριση των βοηθειών θα δίνονται προς τα παραδοσιακά και τα νέα κράτη-μέλη. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Πώς θα ξεβρεθεί σωστή ισορροπία. Γιατί εμείς φοβόμαστε ότι θα βρεθούμε εκτός συναγωνισμού. Όταν ήδη θα έχουν ληφθεί όμως οι αποφάσεις. Θα το μάθουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κάναμε μια ανάκριση και μάλιστα μακροσκελή στον Επίτροπο. Ελπίζουμε ότι θα προλάβει και θα θυμηθεί να δώσει την απάντηση τους σε όλους τους ε, παραμένοντες. Παρακαλώ. Πόσα λεφτά μου δίνετε, Πρόεδρε όσα θέλεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο είναι το περισσότερες ερωτήσεις, αλλά παρακαλώ πολύ καταλάβετε με. Ορισμένα στοιχεία δεν μπορώ να σας τα δώσω, να σας εξηγήσω γιατί. Ε, καταρχήν σε ό,τι αφορά τα θέματα σχετικά με την ανακοίνωση για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ε, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι. Ο καθένας από θα μπορούσε να είναι στη θέση μου ε, αντιπροσωπεύω την ε, Κομισιόν και δεδομένου ότι το κείμενο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Κομισιόν ε, δεν μπορώ να σχολιάσω γιατί αυτό που μετράει δεν είναι οι δικές μου προτάσεις αλλά οι προτάσεις της Κομισιόν. Ελπίζω το τελικό κείμενο που θα βγει από την Κομισιόν να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στις δικές μου προτάσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να μην μπω σε λεπτομέρειες για προτάσεις για τις οποίες θα είμαι εδώ στις 17 Νοεμβρίου το απόγευμα μαζί σας για να τις συζητήσω. Ξέρω, καταλαβαίνω ε, τις ανησυχίες σας, ε, αλλά δεν μπορώ ε, να σας πω τίποτα παραπάνω. Δεύτερον, για την γαλλογερμανική πρόταση. Καλύτερα να καλέσετε τους δύο υπουργούς αν σας ενδιαφέρει αυτή η κοινή πρόταση. Δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω την πρόταση, την θέση του καθενός από τα 27 κράτη-μέλη. Όταν συζητήσει Ισλάμου χώρα στο Συμβούλιο θα έχετε την ευκαιρία να, να δείτε την θέση αυτή. Μπορείτε να συζητήσετε με το Συμβούλιο και στο πλαίσιο της συναπόφασης. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω δημοσίως θέσεις κρατών μελών που εκφράζονται στο Συμβούλιο. Είναι βέβαια πολύ θετικό που τα κράτη-μέλη ασχολούνται, το συζητάνε μεταξύ τους, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω τη θέση τους παρόλο ότι η Γαλλία και η Γερμανία είναι πολύ σημαντικά κράτη-μέλη και η θέση τους σίγουρα θα βαρύνει στην διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν όμως άλλα και άλλα 25 κράτη-μέλη. Μετά μου θέσατε πολλές ερωτήσεις που δεν αφορούν το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Έχουν σχέση με τον Επιτρόπο Παλή. Για παράδειγμα, γενετικά τροπημένες ουσίες, ε, ε, μεταφορά, ταυτοποίηση, ε, ευζοία. Όλα αυτά δεν αφορούν το δικό μου χαρτοφυλάκιο. Τώρα, για το εμπόριο. Έχει σχέση με τις δικές μου αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά το γεωργικό εμπόριο. Για το Μερκοσούρ δεν ξέρω τι δήλωσε ο ε, συνάδελφος Ντεγκούκτ στην Αργεντινή. Ε, εγώ έχω πει καθαρά ότι όσο δεν υπάρχει αξιολόγηση αντικτύπου τύπου επαρκή δεν μπορώ να υποβάλω προτάσεις. Ελπίζω θα την έχουμε το τέλος του χρόνου και μέχρι, και μέχρι τότε και μάλλον όταν τη λάβω θα υποβάλω προτάσεις που θα ενταχθούν στην εντολή που έχει η διαπραγματευτική εντολή που έχει η Κομισιόν. Δεν θα κάνω καμία πρόταση, δεν θα κάνω καμία υπόσχεση προς το παρόν. Ήμουν ως τώρα διαφανής, θα είμαι και από εδώ και πέρα διαφανής. Η Κομισιόν έχει διαπραγματευτική εντολή, λαμβάνουν χώρα διαπραγματεύσεις, εμπιστευτείτε με. Ακόμα και αν το άνοιγμα των αγορών μπορεί να είναι ωφέλιμο για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φτάσουμε μόνο μέχρι το σημείο στο, στο οποίο δεν θα θυσιαστούν επενδύσεις που έχουν γίνει από Ευρωπαίους για τη βελτίωση ποιότητας των δικών τους προϊόντων. Ε, για την ποιότητα ιδιαίτερως έχω μια κόκκινη γραμμή, θα την διατηρήσω. Μέχρι τώρα δεν έχω κάνει καμία πρόταση για το Μερκοσούρ. Για τον Καναδά τα πράγματα δεν προχωράνε πολύ, δεν έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που ανέλαβα εγώ. Ο Καναδάς ε, επίσης είναι συγκρατημένος και εκεί υπάρχουν θέματα ποιότητας, γεωγραφικών ενδείξεων, το γάλα. Όσο δεν υποχωρούν οι Καναδοί δεν βλέπω γιατί θα υποχωρήσουμε εμείς. Μετά αναφέρατε και το Μαρόκο. Το Μαρόκο το διαπραγματεύτηκε η προηγούμενη Κομισιόν. Νομίζω ότι θα επικυρωθεί σύντομα στο Κοινοβούλιο η συμφωνία αυτή. Όπως σας είπα, τη διαπραγματεύτηκε αυτή η συμφωνία η προηγούμενη Κομισιόν και σίγουρα δεν προβλέπει πλήρη απελευθέρωση. Ακόμα και για τις ντομάτες και τα προκυπευτικά ε, δεν προβλέπεται πλήρης, ε, πλήρης άνοιγμα. Υπάρχουν συστήματα ασφάλειας, υπάρχουν ρήτρες ασφάλειας που μας επιτρέπουν να παρέμβουμε όταν δημιουργούνται προβλήματα όπως την ντομάτα. Τώρα, να διατρέξω εντάχει τα διάφορα ζητήματα. Για την κοινή επιστολή ήδη είπα ποια είναι η, απάντησή μου. Μου λέτε, γιατί ενημέρωσα τον τύπο και όχι το κοινοβούλιο. Καταρχήν δεν ενημέρωσα το κοινοβούλιο. Η επιστολή αυτή δεν απεστάλλει στον τύπο, διέρευσε. Είναι μια εσωτερική επιστολή που οι τέσσερις επίτροποι έστειλαν στον πρόεδρο της Κομισιόν. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για αυτό το θέμα στην Κομισιόν. Είναι μια πρόταση των τεσσάρων επιτρόπων στον πρόεδρο της Κομισιόν. Το διευκρινίζω γιατί έγινε διαρροή. Δεν ενημέρωσα, εσάς δεν ενημέρωσα τον τύπο πριν ενημέρωσω εσά. Πρόκειται για μια εσωτερική συνένεση στην, εντός της Κομισιόν και θα τη συζητήσουμε θα συζητήσουμε τι θα περιλαμβάνει αυτό το στρατηγικό πλαίσιο. Είναι στρατηγικό πλαίσιο ε, με τεσσάρων επιτρόπων που έχουν διαφορετικούς προϋπολογισμούς, διαφορετικά, διαφορετικές αρμοδιότητες, αλλά στην εφαρμογή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη διαφάνεια, έτσι ώστε ε, με σεβασμό των στόχων των προϋπολογισμών κλπ. Οι περιοχές στις οποίες ε, εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα να, να καταφέρουν να συντονίσουν καλύτερα την εφαρμογή. Πρόκειται για στρατηγικό πλαίσιο ε, εφαρμογής ο, σε κάθε προϋπολογισμό υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο εφαρμογή που δίνουμε οδηγίες στα κράτη-μέλη για το πώ θα εφαρμόσουν κάθε πρόγραμμα. Και ακόμα και κάθε κράτος μέλος προσπαθεί να συντονίσει τα διάφορα υπουργεία, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, περιφερειακή Ανάπτυξης κλπ. έτσι ώστε να μην αλληλεπικαλύπτονται και να μην αφήνουν εκτό σημαντικά πράγματα αυτό το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να διευκολύνουμε τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη. Θα το ξανασυζητήσουμε όταν μιλήσουμε για το νομοθετικό πακέτο για αυτό το ζήτημα. Για τους ε, κανόνε αγοράς για το γάλα. Το πακέτο γάλα. Οι προτάσει μας θα ζητούν ενίσχυση των ανάσων παραγωγών, υπογραφή συμβάσεων, διαπαγγελματικέ σχέσει και διαφάνεια υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν προκύψει από την ομάδα ε, υψηλού επίπεδου που θα τα δούμε στο πακέτο για την μεταρρύθμιση ΣΚΑΠ. Ε, διαχείριση κρίσεων και εργαλεία, για παράδειγμα, και εδώ απαντώ και σε άλλη μια ερώτηση σχετικά με τα εργαλεία παρέμβαση και διαχείριση κρίσεων. Ε, ναι, θα διατηρήσω το εργαλείο της παρέμβασης, αλλά ως δίχτυ ασφαλείας για τα σιτηρά, το γάλα και κάποια άλλα προϊόντα ασφαλώς και θα διατηρήσουμε την παρέμβαση ως δίχτυ ασφαλείας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην αγορά σιτηρών, το είπα και χτες στο Συμβούλιο Γεωργίας, παρακολουθούμε από κοντά τις τιμές. Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν έχουμε κάποια μαγική ράβδο, δεν μου έχουν κληροδοτήσει μια τέτοια μαγική ράβδο η προκατοχή μου. Ε, ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας θα τα χρησιμοποιήσουμε συμπεριλαμβανομένης και της διάθεσης αποθεμάτων που διατηρούμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τεράστιες οι ποσότητες αυτές, αλλά αυτές που έχουμε θα προσπαθήσουμε να τις ε, διακινήσουμε στην αγορά μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα έχουμε σαφή εικόνα της παραγωγής, της σοδιάς δηλαδή, της φετινής χρονιάς. Αυτό θα πρέπει να γίνει πριν διαθέσουμε τα αποθέματά μας στην αγορά και το είπα και στο Συμβούλιο, βλέπουμε μια αύξηση τιμής και που ενδεχομένως επηρεάζεται από τις αποφάσεις της Ουκρανίας. Όμως η παραγωγή δεν βρίσκεται στα επίπεδα που ήταν 2007-2008, είναι κοντά στο μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Συνεπώς ε, γενικά δεν υπάρχει έλλειψη σιτηρών. Και μου, αναφ- κάνετε και μια ερώτηση για την κερδοσκοπία ε, και τις μεγάλες διακοιμάσεις τιμών. Ε, μαζί με τον Επίτροπο Εσωτερική Αγορά, τον κύριο Μισελ Μπαρνιέ, επενέβημεν μαζί, παρενέβημεν μαζί λοιπόν, για να ζητήσουμε ρύθμιση των, της Αγοράσει το μεταποιημένο προϊόντο για να ε, αποφύγουμε την κερδοσκοπία και να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Ε, συμφωνώ και θα ήθελα να γίνει το ίδιο και για τα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε λίγη τάξη δηλαδή ε, στο πώς γίνονται οι αγορές και οι πωλήσει, οι αγοροπολισίες στις αγορές και να αποφύγουμε κερδοσκοπίες σε ό,τι το νομοθετικό πακέτο και το χρονοδιάγραμμα. Ο κ. Λάιον είπε ότι ε, βλέπει πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα. Σωστό, είναι πολύ φορτωμένο, αλλά δεν λαμβάνουν χώρα τα πάντα την ίδια χρονική στιγμή. Έχουμε μέχρι το τέλο του χρόνου το πακέτο για το γάλα και του χρόνου ελπίζω θα έχουμε μια τελική απόφαση να υιοθετηθεί αυτό το πακέτο. Το νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση ΚΑΠ θα φτάσει τον επόμενο Ιούλιο. Ε, αυτή τη στιγμή ε, προετοιμάζουμε την ανακοίνωση με τις ε, γενικές γραμμές προσανατολισμού. Μετά θα ξεκινήσουν τη διαβούλευση, αλλά επί τη βάση εγγράφου προσανατολισμού της Κομισιόν. Ε, μετά από αυτή τη συζήτηση θα λάβω υπόψη όλες τις παρατηρήσεις που εσείς θα κάνετε, θα κάνετε το Συμβούλιο κλπ για να προετοιμάσω το νομοθετικό πακέτο που, επαναλαμβάνω, θα είναι έτοιμο τον Ιούλιο. Για τι εφαρμοστικέ πράξει, για τι εκτελεστικές πράξεις, ε, είπα στου συντονιστέ τη ε, ε, ε Επιτροπή ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό. Για την στρατηγική προσέγγιση για τον προπολογισμό και σχετικά με τη μετάρρυνση ΚΑΠ, για τον προπολογισμό υπάρχει χρονοδιάγραμμα που νομίζω το παρουσίασε ο πρόεδρος της ε, Κομισιόν στην ομιλία του στο Κοινοβούλιο. Αυτό μπορώ να σας πω, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι σε πρώτη φάση θα γίνει η ενδιάμεση αναθεώρηση και μετά θα εκδοθεί ανακοίνωση. Επίσης θα γίνει του χρόνου η νομοθετική παρουσίαση, νομίζω την Άνοιξη και βέβαια αμέσως μετά το νομοθετικό πακέτο για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό το νομοθετικό πακέτο για να δώσουμε μια ε, εικόνα στους παραγωγούς για το τι θα γίνει μετά το 2014. Μέχρι τώρα η νομοθεσία μας φτάνει μέχρι το 2013. Θα πρέπει να δώσουμε μια προοπτική για την περίοδο μετά το 2014 στους παραγωγούς και στους αγρότες. Απάντησα στον κύριο Νίκολσον για το θέμα του ότι ο τύπος ενημερώνει πριν να ενημερώσει ο Επίτροπος. Δεν είναι εδώ βέβαια ο κ. Νίκολσον, αλλά επαναλαμβάνω, κάθε φορά που μου το ζητάτε ή κάθε φορά που νομίζω ότι χρειάζεται, ε, έρχομαι εδώ ε, και σας ενημερώνω. Αυτό που διέρευσε ήταν κάτι εσωτερικό της Κομισιόν. Κ. Χόισλινγκ, ασφαλώς και θα συνεχίσουμε την δημόσια διαβούλευση, θα κάνουμε δημόσια διαβούλευση επί τη βάση της ανακοίνωσης. Έκθεση Μποβέ και συνέχεια που θα δοθεί. Ασφαλώς κάποια πράγματα θα συμπεριληφθούν στο νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ζήτησα από την υπηρεσία μου να αναλύσουν τις προτάσεις, να δουν τι μπορούμε να συμπεριλάβουμε. Υπάρχουν όμως και κάποια στοιχεία τα οποία δεν εξαρτώνται από μένα ή μόνο από μένα έχουν σχέση με την ε, βιομηχανική πολιτική ε, για τον τομέα της βιομηχανίας των τροφίμων. Υπάρχει μια ομάδα υψηλού επίπεδου για την ε, αγροτροφημική αλυσίδα. Ε, κάποιες άλλες προτάσεις έχουν σχέση με, την, με τον ανταγωνισμό. Αφού τις αναλύσουμε θα συζητήσω και με τους συναδέλφους μου να δω πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη και τα θέματα τη αλυσίδα και τα θέματα του ανταγωνισμού και πού δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα δική μου. Εκφεύγουν των αρμοδιότητων μου. Για το θέμα της ποιότητας, του πακέτου ποιότητας, θα υποβληθούν προτάσεις για την ε, σήμανση που θα περιλαμβάνει το τόπο παρασκευής. Ιδιαίτερως για συγκεκριμένα τοπικά προϊόντα, ή προϊόντα από ορεινές περιοχές. Θα το δούμε. Για την κοινή επιστολή πώς θα εφαρμοστεί. Θα το δούμε όταν είναι έτοιμη η πρόταση κυρία Γέγκλε. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα την, τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της επιστολής. Για τα σιτηρά απάντησα. Για την ανάπτυξη της υπαίθρου επίσης ετέθησαν διάφορα ερωτήματα, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ΚΑΠ. Διαθέτει ένα σημαντικό προπολογισμό και θα προσπαθήσουμε με τις προτάσεις μας να λάβουμε υπόψη και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας αλλά και την εξέλιξη των τοπικών προϊόντων, των μικρών ε, μονάδων παραγωγής, την καινοτομία, ε, τις πωλήσει εγκύτητος κλπ. Αλλά αυτό θα το δούμε ε, στο Νοέμβριο όταν ξανάρθω να σας μιλήσω. Πολιτική ανταγωνισμού και κοινή αγροτική πολιτική. δεν σκοπεύω να αλλάξω του κανόνε ανταγωνισμού. Υπάρχει επίτροπο ανταγωνισμού και υπάρχουν κανόνε ανταγωνισμού. Πλην όμω, η συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει τη δυνατότητα ο αγροτικό τομέα να διαθέτει κοινέ οργανώσει αγορά με δικού του κανόνε ανταγωνισμού εξαιτία τη ιδιαιτερότητα του αγροτικού τομέα. <clears throat> Δεν θα ζητήσω άλλε εξαιρέσει πέραν αυτών που περιλαμβάνονται ήδη συνθήκη. Δεν θέλω να επηρεαστεί η συνολική λειτουργία των αγορών. Δεν σκοπεύω δηλαδή να αλλάξω τους κανόνες ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω απλώς οι κανόνες ανταγωνισμού που έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα να τύχουν σεβασμού. Δεν θέλω να μπερδεύουμε τα πράγματα. Έχουμε μια ιδιαιτερότητα ως αγροτικός τομέας και γι' αυτό το λόγο έχουμε κανόνες συνταγωνισμού που ορίζονται από τις κοινέ οργανώσεις αγοράς. Αυτά για να αποφεύγουμε τη σύγχυση και τις παρανοήσεις. Η κυρία Ράνς Γκαρσία. στο πακέτο ποιότητα ε, θα κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα σε γεωγραφικέ ενδείξει και ε, προστατευόμενε ενδείξει προέλευση. Ε, σίγουρα θα το δείτε. Δεν πρόκειται να καταστρέψουμε κάτι που ήδη λειτουργεί. Βέβαια θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το σύστημα να γίνει πιο σαφέ. Αυτό ναι. Οι ονομασίε προέλευση, οι γεωγραφικέ ενδείξεις, η ο ρόλος των επαγγελματικών σωματείων να, ε, θα γίνει πιο σαφής η διάκριση μεταξύ τους κλπ. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα όταν δείτε το πακέτο ποιότητας. Συντονισμός ανάμεσα στην εμπορική και την κοινή αγροτική πολιτική. Κύριε Μαγκίνες δηλαδή. Ε, ξέρω ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Δεν... Μάλλον, ο αγροτροφημικός τομέας είναι ο μεγαλύτερος κλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχει σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε προκειμένου να διατηρήσουμε το αγροτικό μας μοντέλο για το οποίο έχουμε επενδύσει πάρα πολύ. για το γάλα, αν θα αντικατασταθούν οι ποσοστώσεις από τα συμβόλαια ή οι ποσοστώσει θα διατηρηθούν μέχρι το 2015 έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε το 2010 και ελπίζω ότι με απόφαση που θα ληφθεί του χρόνου προτείνουμε συστήματα παράλληλα με τις ποσοστώσεις που θα επιτρέψουν στους παραγωγούς γαλακτός να οργανώσουν καλύτερα την παραγωγή τους, να είναι πιο παρόντες στις αγορές τη στιγμή της διαπραγμάτευσης των τιμών, των ποσοτήτων και της υπογραφής συμβάσεων και θα το δείτε και στο πακέτο το οποίο θα υποβάλω, δεσμεύομαι πριν το τέλος της θητείας μου, οπότε πριν το τέλος των ποσοστώσεων, να υποβάλω έκθεση και αν χρειάζεται να πάρουμε και πρόσθετα μέτρα ή να ενισχύσουμε κάποια μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, να το κάνουμε για να αποφύγουμε την αστάθεια στον ε, τομέα του γάλακτος. Αυτά όμως, ε, μάλλον αυτά που προτείνουμε, θα λειτουργήσουν παράλληλα με το σύστημα των ποσοστώσεων που δεν θα ε, φτάσει το τέλος του πριν το 2015. Για τους νέους ε, γεωργούς. Και Νικολέσκου, ε, λίγη υπομονή. Θα δούμε το θέμα της εγκατάστασης των νέων γεωργών ή των καινούριων γεωργών, γιατί οι καινούριοι γεωργοί δεν είναι πάντοτε νέοι. Το είπα σε ένα συνέδριο νέων γεωργών την περασμένη εβδομάδα ότι αν δεν εξασφαλίσουμε τη δική τους συνειδητοποίηση, ε, τη δική τους ε, εμπιστοσύνη στο μέλλον, έχουμε αποτύχει στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θα υποβάλουμε πρόταση, δηλαδή για το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ε, νέους και καινούριους παραγωγούς να εγκατασταθούν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Θα λάβουμε υπόψη και τις διαφορετικές κατηγορίες γεωργών και τις διαφορές ανάμεσα σε χώρες. για τον προϋπολογισμό, κ. Λεβαντόφσκι. Α, για την... Ε, δεν έχουμε μετάφραση, λέει. Ε. θα προσπαθήσω... Θα προσπαθήσω να τα πω στα αγγλικά. Θυμάμαι ότι ρωτήσατε, το ρωτήσατε αυτό και κατά τη διάρκεια της ακρόασης μου και σας απάντησα. Ε, το θέμα ε, έχει σχέση με την ευζοία των ζώων. Δεν έχει σχέση με μένα. Ο Επίτροπος Νταλή θα απαντήσει. Γιατί αυτός είναι ο υπεύθυνο για τον κανονισμό της ευζοίας. Ευχαριστώ που το διευκρινίσατε. Είναι κάτι πολύ καινούριο για πολλούς από εμά. Δεν νομίζω ότι είναι καινούριο, λέει ο Επίτροπος. Η διάκριση ανάμεσα στα διάφορα χαρτοφυλάκια είναι πολύ σαφής η ασφάλεια των τροφίμων, η ευζοία των ζώων, η προστασία του καταναλωτή ε, ανήκουν στον Επιτρόπο κ. Νταλή. Μια απάντηση γρήγορη. Δε, όλες οι οργανώσεις ε, πίεσης, λόμπι ε, της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου μου ζήτησαν να απευθυνθώ σε εσά. Ε, θα του πω ότι απευθύνονται σε λάθο άνθρωπο. Γι' αυτό μόνο το θέμα, πέστε του ότι απευθύνονται σε λάθο άνθρωπο, εντάξει. Ε, για το θέμα του προπολογισμού. Ε, δεν ξέρω τι εννοεί ο κ. και λέγοντα ότι ε, ο προπολογισμό τη ΚΑΠ θα πρέπει να μειωθεί ω ποσοστό του συνολικού προπολογισμού ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν θα διαφωνούσα υπό την προπόθεση ότι ο συνολικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθεί. Γιατί αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα σχέδιά μα, οι φιλοδοξίε μα για τον αγροτικό τομέα και την αγροτική πολιτική, θα πρέπει το απόλυτο ποσό να παραμείνει. Νομίζω ότι αυτά δεν έχουν να πω τίποτα άλλο. Ε, direct Άμεσες πληρωμές και άλλα θέματα τα σχετικά με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα τα συζητήσουμε όταν ε, υποβάλουμε το, τις προτάσεις μας στην ανακοίνωση 27 Νοεμβρίου. Το είπα από την αρχή. Ε, ναι, ναι, το ξέχασα. Μου ζητάτε να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας. Δεν τις γνωρίζω. Η, Ουγγρική Προεδρία θα σας τις παρουσιάσει. Η μικρή ε, Γεωργή ε, θα δείτε στις 17 Νοεμβρίου θα υποβάλω μια ανακοίνωση και εκεί ε, κάνουμε αναφορές στην γεωργία μικρών παραγωγών και το πώς μπορούμε να προωθήσουμε την παραγωγή τους. Θα τα δείτε αυτά στις προτάσεις που θα κάνω. Σας ευχαριστούμε κύριε πίτροπε Άρζαν για αυτό το μακροσκελέστατο ερωτηματολόγιο αλλά θα πρέπει να διοργανωθούμε ίσως και διαφορετικά. Είμαστε σε μια φάση εντατικών εργασιών το πρόγραμμα που μα παρουσιάσατε ήδη εσεί ήταν πλουσιότατο. Έχουμε νομοθετικά πακέτα. Θα πρέπει να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε το μέλλον τη ΚΑΠ. Θα πρέπει ίσω να πολλαπλασιάσουμε τι συναντήσει μα, να έρχεστε κι εσεί πιο συχνά να συναντάτε τα μέλη τη Επιτροπή μα και εμεί να διοργανώσουμε καλύτερα τι δικέ μα τι εργασίε. Δεν μπορούμε να περνάμε ένα ολόκληρο απόγευμα να ρωτάμε ό,τι μας περνάει από το μυαλό. Πρέπει να επικεντρωθούμε στα μεγάλα ζητήματα, μεγάλα ερωτήματα και να ζητούμε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον Επίτροπο. Και ο Επίτροπος προφανώς θα μας δίνει τη δική του την άποψη. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εμείς νομοθέτες. Δεν είμαστε πλέον ένα κοινοβούλιο που απλώς αποφαίνεται για μια έκθεση, μια γνωμοδότηση. Η τελική ευθύνη θα είναι μοιρασμένη και σε εμά. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να διαχειριστούμε σωστά την ευθύνη που μα αναλογεί. Όχι απλώς να ζητούμε και να ρωτούμε, αλλά να κάνουμε και προτάσεις και να τις επεξεργαζόμαστε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Τσόλος, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ένα λεπτό διακοπή και συνεχίζουμε ευθύ αμέσω με το workshop. Possiamo iniziare? Να ξεκινήσουμε. Elisabeth Jägel là. Per favore, prendete posto. Η κυρία Γέγκλε είναι μαζί μας. Καθίστε παρακαλώ. Το Department B, vedo tutti che chiacchierano. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλά πηγαδάκια. Allora iniziamo col punto Ξεκινάμε με το σημείο 5 λοιπόν της σημερινή συζήτησης, ρόλος των γυναικών στη Γεωργία και στις περιοχές της Επέθρου. Ξεκινάμε με αυτό το πολύ σημαντικό σεμινάριο εργαστήριο. Πρώτα απ' όλα, εξ ονόματος ολόκληρης της Επιτροπής μας, να καλωσορίσω τους ε, προσκεκλισμένους μας. Κυρία Σέλι Σόρταλ του Πανεπιστημίου Queen στο Belfast και την κυρία Μπετίνα Μποκ του Πανεπιστημίου του Βαντενίγκε. Όπως θα ξέρετε, η Επιτροπή μας θα καταρτήσει μια γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για το ρόλο των γυναικών στη γεωργία στις περιοχές της Πέθου. Για αυτό το θέμα έχει αναλάβει η συνάδελφος, η κυρία Γέγκλε. Η θέση και η συνεισφορά των γυναικών στο τομέα αυτό και στις εν λόγω περιοχές έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Όμως αυτή η ανάπτυξη καλύπτει πολλές ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Με αυτό το εργαστήριο λοιπόν θέλουμε να εμβαθύνουμε την, και να δούμε το εργασιακό προφίλ των γυναικών στον τομέα της γεωργίας. Ευθύ αμέσω θα δώσω το λόγο στις προσκεκλημένες μας, εκτός αν θέλει να παρέμβει πρώτη η κυρία Γέγκλε. Απευθείας λοιπόν θα ακούσουμε τις προσκεκλημένες, η κυρία Μποκ και μετά η κυρία Σόρταν. Θα μας παρουσιάσουν τα πορίσματα του έργου τους. thank you very much for the invitation uh, to present these presentations. I think both Bettina and I have found it very interesting. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσκλησία σας να παρουσιάσω τα πορίσματα του έργου μας. Και εγώ και η Μπετίνα έχουμε μια μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίσουμε. Λέγομαι Σάλι Σόρταλ και θα ξεκινήσω μιλώντας για το ρόλο των γυναικών στην ε, Γεωργία σε όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ήδη αργά και ότι είσαστε κουρασμένοι. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να είμαστε σύντομες. Μου ζητήθηκε συγκεκριμένα να μιλήσω για τις διαφορές του των ρόλων που έχουν οι γυναίκες στη Γεωργία από άποψη νομικού και πολιτικού πλαισίου και να διατυπώσω κάποιες συστάσεις για την περίοδο μετά το 2013 για να βελτιωθεί η προσώπηση των φύλων στα πλαίσια της ΚΑΠ. Ε, περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε και στο έγγραφο που θα βρείτε μπροστά σας και σε αυτή την παρουσίαση θα επικεντρωθώ πολύ σύντομα στην θέση των γυναικών στη Γεωργία, να δούμε ποιο είναι το εργατικό δυναμικό που σχηματίζουν οι γυναίκες, ποιες είναι οι στενές του διασυνδέσεις. Με την έρευνα που κάναμε εγώ και η Μπετίνα Μποκ και θα δούμε κάποια στοιχεία για το πώς έχουν πρόσβαση στη γη οι γυναίκες και τι γίνεται με τις γυναίκες συζύγους στις εκμεταλλεύσεις, καθώς αυτές είναι η πλειοψηφία των ε, γυναικών που αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Οι νέε αφήξει λοιπόν στη Γεωργία θα μας απασχολήσουν, καθώς και το πολιτικό και νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες συστάσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν κάποια προκαταρτικά, προειδοποιητικά μάλιστα σχόλια. Θα γνωρίζετε όλοι ότι υπάρχουν σοβαρές ε, ανά την Ευρώπη ως προς την μορφή γεωργία, τι καλλιέργειες δηλαδή και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με τι γυναίκε και τη γεωργία. Ο ρόλο των γυναικών στη γεωργία εξαρτάται από το μέγεθο και το είδο τη καλλιέργεια. και πολλέ φορέ και από τι τοπικέ αγορέ η την μορφη τη υπαιθρου οι σημαντικότερε διαφορέ εντοπιζονται μεταξυ παλιων και νεων κρατων μελων βεβαίω. η κατάσταση των γυναικών έχει δυσκολέψει λίγο εξαιτία των συγκρίσιμων δεδομένων που δεν διαθέτουμε ώστε να κάνουμε συγκριτική μελέτη. Όμως, το ζήτημα αυτό ίσως να το επιλύσουμε με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο μετά το 2013. Αυτή είναι μια φωτογραφία που μου επέτρεψε να χρησιμοποιήσω μια τοπική εφημερίδα Ιρλανδών γεωργών του πολίτε στην ε, Βόρεια Ιρλανδία. Ο λόγος που σας δείχνω τη φωτογραφία αυτή είναι για να δείτε ότι στη φωτογραφία υπάρχει μία και μόνο γυναίκα και αν χρησιμοποιήσετε ένα μεγεθυντικό φακό όπου θα δείτε στο φόρουμ αυτό να υπάρχει το πολύ άλλη μια γυναίκα. Αν τα καταφέρετε να βρείτε κι άλλη, θα σα δώσουμε και βραβείο. Αυτό δείχνει πόσο περιορισμένο είναι ο ρόλο των γυναικών στη Γεωργία ή τουλάχιστον η εκπροσώπησή του και είναι ένα ανδροκρατούμενο σαφέστατα τομέα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, συμβολή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό της Γεωργίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι συμβάλλουν σημαντικότατα σε αυτό το εργατικό δυναμικό και τις ε, ε, τι γεωργικέ δραστηριότητε. Το 41% του εργασιακού δυναμικού στη γεωργία είναι γυναίκε. Υπάρχει διαφορά βέβαια μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Τι περισσότερε φορέ εκμεταλλεύσει ξεκινάνε σε οικογενειακό επίπεδο και τι περισσότερε γεωργικέ δραστηριότητε τι ε, διεκπεραιώνει η οικογένεια. Υπάρχουν φυσικά διαφορέ μεταξύ των κρατών τη Ευρώπη και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στα νέα κράτη-μέλη από την πλευρά των γυναικών. Αυτό τίνει να συσχετίζεται με την διάρθρωση της γεωργίας και της οικονομίας στα νέα κράτη-μέλη. Δεν είναι απλώς ένα θέμα ισότητας των φύλων. Είναι πιο πολύπλοκη η εξήγηση. Τα στατιστικά τώρα στοιχεία μας δίνουν ε, περιορισμένες δυνατότητες κατανόησης τη συμβολή των γυναικών στις γεωργικές δραστηριότητε. Ε, Ποιοτικέ έρευνε, μελέτε έδειξαν ότι οι στατιστικέ τελικά υποτιμούν και υποβαθμίζουν το ε, ρόλο των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, διότι πολλές φορές δεν αντικατοπτρίζεται το έργο τους ε, μέσα στις μέρες και τις εβδομάδες. Ε, κάποιες βοηθητικές εργασίες που μπορεί να μπερδεύονται με τα όσα κάνουν στον οικοκυριό τους στα πλαίσια της γεωργικής εκμετάλλευσης. Με αυτόν τον πίνακα δίνουμε κάποια εικόνα μερικών χωρών και τη σύγκριση για το πώς εκπροσωπούνται γυναίκες και άντρες ε, στο εργατικό δυναμικό μεταξύ παλαιών και νέων κρατών μελών. Βλέπουμε πόσο υψηλά είναι τα ποσοστά στη Λιθουανία και Λετωνία και πόσο χαμηλά στην Ιρλανδία και τη Δανία. Πάντω, ένα από τα ερωτήματα που θα πρέπει να θέσουμε στου εαυτού μα είναι να σκεφτούμε εάν η τάση αυτή είναι θετική ή εάν εκπροσωπεί γενικότερε τάσει ισότητα των φίλων στη Γεωργία ή όχι. Ένα από τα στοιχεία που σχετίζονται με την ε, ε, ΚΑΠ είναι η διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και πώς αυτό επηρεάζει τα εισοδήματα. Τα συγκρίσιμα δεδομένα μας είναι ελάχιστα. Όμως οι εθνικές μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να δραστηριοποιούνται και σε αυτό το τομέα, το τομέα διαφοροποίησης των γεωργικών ε, δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλέ εξηγήσει γι' αυτό. Σε πολλέ περιοχέ τη Ευρώπη οι γυναίκε που απασχολούνται στη γεωργία έχουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλύτερα προετοιμασμένες για να αναλάβουν επιχειρησιακές δραστηριότητες, να αναπτύξουν στρατηγική σκέψη. Είναι επικεντρωμένε επίση στην ε, ανατροφή των παιδιών του ε, στι γεωργικέ του αρμοδιότητε κάποιε φορέ. Η Μπετίνα με την έρευνά τη έδειξε ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση οι γυναίκε στην διαφοροποίηση το γεωργική και ενδιαφέρονται περισσότερο στο να αναπτύξουν για το να αναπτύξουν πρωτοβουλίε που χρειάζονται πιο βραδία εκταμείευση κεφαλαίου. Αυτό όμω διευκολύνει τη διαφοροποίηση και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν θα καταλέξουμε στι συστάσει. Επίση, κάποιε ιδιαίτερε ενδείξει για τα νέα κράτη-μέλη υπάρχουν εδώ. Όπω έδειξε η ερευνά μα, δεν υπήρχε πάντοτε η απαραίτητη υποδομή προκειμένου οι πρωτοβουλίες διαφοροποίησης γεωργικής να υλοποιηθούν. Κάποιες φορές επίσης οι πρωτοβουλίες για του είδους αυτού τη διαφοροποίηση απαιτούν και κάποιες κεφαλογικές επενδύσεις. Οπότε και αυτό μπορεί να είναι ένας παράγοντας εργασία των γυναικών ε, σε μια γεωργική εκμετάλλευση είναι πολύ σημαντική για την επιβίωση την ίδια του αγροκτήματο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε. Η καθιερωμένη τάση είναι οι γυναίκες που βρίσκονται σε εκμεταλλεύσεις συχνά όλο και περισσότερο να ε, δουλεύουν εκτός αυτό είναι μια επιλογή ζωή. Πολλέ φορέ οι γυναίκε επιλέγουν να ακολουθήσουν τη δική του σταδιοδρομία, αλλά αυτό εξαρτάται και από την περιφέρεια και την περιοχή, ανάλογα με το μορφή τη εκμετάλλευση, την δομή τη, την ε, όλη κουλτούρα και τι ευκαιρίε που υπάρχουν στην τοπική αγορά Κάποιε φορέ η εμπλοκή των γυναικών στη Γεωργία μπορεί να σημαίνει και ένα αδιέξοδο, έλλειψη άλλη επιλογή. Υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές ε, ανησυχίες από πλευράς των γυναικών και οικονομικού ε, περιεχομένου πρωτοβουλίες προκειμένου να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης και, να, και νέες πηγές εισοδημάτων. Τώρα, για την σύγκριση γυναικών και ανδρών και πώς λειτουργούν ανάλογα με τις επιλογές που έχει κάνει ο σύντροφός τους. Βλέπουμε ότι επηρεάζονται εδώ οι στρατηγικές της γεωργικής εκμετάλλευσης ανάλογα με αυτή την ισορροπία. Ένα από τα θέματα που έχει πρωταρχική σημασία είναι πώς ε, έχουν πρόσβαση οι γεωργοί στη γη. Διότι η γεωργία δεν είναι μια οποιαδήποτε δραστηριότητα. Δεν μπορεί κανείς να εκπαιδευτεί και να αρχίσει να αγωνίζεται για να βρει μια θέση εργασία στην ε, αγορά. Πρέπει να έχει ένα κομμάτι γης, το οποίο είτε θα κληρονομήσει θα έχει πρόσβαση σε ένα νέο ε, τεμάχιο γης. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερες ικανότητες. Ένας από τους βασικούς παράγοντες λοιπόν που καθορίζει την μεταβίβαση των αγροτοτεμαχίων είναι οικονομικός, οικονομική βιωσιμότητα όμως της βιομηχανίας εξαρτάται από το αν η γη μεταφέρεται κατά τρόπο ώστε να μένει ακέραιο το αγροτεμάχιο. Υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα νομικών πλαισίων ανά την Ευρώπη που καλύπτουν ακριβώς το σημείο αυτό, τη μεταφορά, τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της γης. Από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο που μπορεί κανείς να αφήσει σε ένα κλειονόμο τη γη του, μέχρι τη Δανία που πρέπει να αγοραστεί το κομμάτι γης. Ή τη Γαλλία και τη Γερμανία όπου υπάρχει κοινή ιδιοκτησία για το ζευγάρι ή την Νορβηγία όπου το μεγαλύτερο παιδί είναι ο νόμιμος κληρονόμος. Μεγάλη λοιπόν νομική ποικιλία και μεγάλο φάσμα νομικών πλαισίων. Βεβαίως, το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τη γεωργία και ιδίω από την πλευρά των γεωργών εξαρτάται και από την κουλτούρα του κάθε μέρου. Οι άντρε είναι συνήθω ιδιοκτήτε και υπεύθυνοι του γατομαχίου. Από το 2007 έχουμε δεδομένα που δείχνουν ότι 78% των γυναικών ε, στα αγροκτήματα είναι σύζυγοι. Τώρα, ιδιοκτήτε αγροτεμαχίων, ε, γυναίκε, ε, βλέπουμε στοιχεία για την Ευρώπη των 27. Στις πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις συνήθως είναι ιδιοκτήτριες οι γυναίκες. Και ιδίω αν η γεωργική επασχόληση είναι μερικής, μερικού χρόνου. Τώρα, το θέμα είναι αν όλα αυτά εκπροσωπούν και τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Και το πώς αλλάζουν τα πράγματα στα νέα κράτη-μέλη είναι σημαντικό, διότι δεδομένη της υψηλής αναλογίας των υψηλών ποσοστών γυναικών που είναι κάτοχοι και ιδιοκτήτε των αγροτεμαχίων που είναι ιδιαίτερα μικρά, εδώ προκύπτουν και πολλέ ε, συνέπειε που θα επηρεάσουν το μέλλον τη ΚΑΠ για το 2013 και μετά. Για το τι θα γίνει επίσης με, τα μεγάλα, με τις μεγάλες ε, εκμεταλλεύσεις. Βλέπουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η εκμετάλλευση, τόσο λιγότερες ιδιοκτήτριες γυναίκες και κάτοχοι γυναίκες υπάρχουν. Και τούμπαλιν. Τώρα, οι πληρωμέ τη ΚΑΠ είναι σημαντικό να πούμε ότι πηγαίνουν προ τον κάτοχο, τον ιδιοκτήτη του αγροτομαχίου. Οπότε, ενώ η εκπαίδευση στοχεύει τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του, τελικά οι σύζυγοι δεν συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Αυτό να είναι να είναι και απλό να ε, αντιμετωπιστεί. Στι γεωργικέ επίση οργανώσει συνήθω κυριαρχούν οι άντρε. Στι εθνικέ επιτροπέ για την κατάρτιση προγραμμάτων, τι γεωργικέ δηλαδή οργανώσει, ε, τα μέλη τείνουν να είναι αποκλειστικά και μόνο άντρε. Η πλειοψηφία των ε, γυναικών στι εκμεταλλεύσει έχουν λοιπόν κατηγοριοποιηθεί ω σύζυγοι. Κάποιε φορές οι σύζυγοι αυτοί ασχολούνται ακριβώς με τη διαχείριση των εκμεταλλεύσεων και με τη λήψη των αποφάσεων και με πρακτικές εργασίες κάποιες φορές, όπως αυτό που είπαμε για τη διαφοροποίηση. Από την πλευρά της πολιτικής όμως είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύσουμε και αυτές τις συζύγους. Κάποιοι μιλάνε για τους νεοαφιχθέντε, τι νέε αφήξει στον ε, χώρο τη Γεωργίας. Η ε, Eurostat δεν μου έδωσε συγκεκριμένα στατιστικά λεπτομερή στοιχεία για τις νέες αφήξεις στην ε, Γεωργία. Όμως, ε, έχουμε αναλάβει μέτρα για να διευκολύνουμε αυτές τις νέες αφήξεις. Η Σουηδία και η Ισπανία έδωσαν επιπλέον κίνητρα, εάν οι νεοαφιχθέντες ήταν γυναίκες. Δεν ξέρουμε όμως εάν αυτό προωθεί την ισότητα των φύλων, ούτε ακριβώς ποιοι είναι νεοαφιχθέντες δεν ξέρουμε αν βελτιώνεται η οικονομική βιωσιμότητα μια γεωργική εκμετάλλευση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να τα αποδεικνύουν. Δεν ξέρουμε επίση αν στρέφεται η λειτουργία μια εκμετάλλευση προ περιβαλλοντικά φιλικότερε μεθόδου. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον η συμμετοχή των γυναικών ε, συνάδει και με του μελλοντικού στόχου τη ΚΑΠ. Αλλά αυτό δεν ξέρουμε αν επηρεάζεται από το γεγονό ότι οι γυναίκε ε, τείνουν να είναι ιδιοκτήτριε σε μικρότερε εκμεταλλεύσει και αν συμβιβάζεται με τι σύγχρονε τάσει τη αγορά. Πάντω υπάρχουν κάποιε γυναίκε στι νέε αφήξει στην αγορά τη Γεωργία, στην Νορβηγία και σε άλλα κράτη. Δεν ξέρουμε γιατί όμω και αν είναι μια θετική τάση. Ω προ το νομικό και πολιτικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν σχετικοί κανονισμοί. Αλλά υπάρχουν περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία για το πόσο αποτελεσματικοί έχουν υπάρξει ω τώρα με ένα από τα βασικότερα ζητήματα που ανακοίτει και από προηγούμενα έγγραφα που μελέτησα είναι ότι ο κάτοχο και ιδιοκτήτη, εφόσον είναι άντρα, τίνει να λαμβάνει τη στήριξη τη άμεση πληρωμή και το καθεξή. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πούμε πώ αυτό μπορεί να αλλάξει, να μεταστραφεί και με ποιο σκοπό. Ε, αν μιλάμε για εισόδημα και όχι κέρδο. Και επίση το θέμα είναι πώ θα επιληθεί από την άποψη των φίλων το ζήτημα τη ιδιοκτησία τη γη. Η διαφοροποίηση, η κατάρτιση, η συμμετοχή των γυναικών είναι θέματα όπου υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να επιφέρουμε βελτιώσεις. Ω προ την οδηγία για την ίση μεταχείριση των συζύγων και των αυτοαποσχολούμενων εργαζομένων, είναι η 8-20-10-41 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντική ε, νομοθετική πράξη για το ρόλο των ε, νεαρών γυναικών συζύγων. Ε, σκοπό έχει να συνδράμε τις σύζυγους και στη μετρότητα και από την άποψη της κοινωνική προστασίας εφόσον είναι εργαζόμενες. Τα κράτη-μέλη είχαν δύο χρόνια για να υλοποιήσουν την οδηγία αυτή στη διάθεσή τους και μου ζητήθηκε να δω σε τι θέση βρίσκονται οι νεαρές γεωργοί που είναι αφιχθείς στο τομέα της γεωργίας. Κοίταξα κατά πόσον υπάρχουν κίνητρα για να αυξηθούν οι αριθμοί των γυναικών αυτών και γιατί, γιατί να αποτελεί αυτό στόχο. Αυτό ήταν το ζήτημα. Η Μπετίνα Μποκ θα μιλήσει για την σημασία της περιφερειακής και αγροτικής αγοράς για τις γυναίκες. Ξέρουμε από τα παλιά και τα νέα κράτη-μέλη πάντως ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες πιθανότητες να, να φύγουν από τις περιοχές της υπαίθρου για σκοπούς απασχόλησης. Ε, σημασία έχει κατά πόσο οι γυναίκε μπορούν να παραμείνουν στην εκμετάλλευση και να έχουν και πρόσβαση στι γεωργικέ δραστηριότητε προκειμένου να απασχοληθούν ω εργαζόμενε. Υπάρχουν κάποιε αποδείξει ότι προγαμιαίε συμφωνίε αυξάνονται συνεχώ στι ε, γυναίκε να μην προβάλλουν αξιώσει λόγου χάρη οι σε περίπτωση διαζυγίου ή να μην επηρεάσουν την οικονομική βιωσιμότητα τη εκμετάλλευση. Ε, σε περίπτωση που είναι αυτοαποσχολούμενε εργαζόμενε οι γυναίκε και το εισόδημά του συμβάλλει στην ε, βελτίωση λειτουργία τη εκμετάλλευση, πρέπει αυτό να αποδεικνύεται. Και <clears throat> θα πρέπει βεβαίω να εξασφαλίσουμε και τα οικονομικά δικαιώματα αυτών των γυναικών. Κάποιε συστάσει τώρα για μετά το 2013. Πρώτα απ' όλα, Υπάρχουν κάποια συνολικά δεδομένα τα οποία δεν έχουν ακόμη μελετηθεί πλήρως και υπάρχουν και πολλές ελλείψεις φυσικά. Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε κάποια από τα ζητήματα για των μελετών σχετικά με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να μελετήσουμε καλά τη διάρθρωση της ε, γεωργίας όσο έχει σήμερα και επίσης να ζητήσουμε περισσότερες, ε, περισσότερη ανάλυση των υπαρχόντων δεδομένων. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα συμβίλημα στατιστικών δεδομένων που να καταγράφει κατά λεπτό στην κατάσταση των γενικών στι γεωργικέ εκμεταλλεύσει, πώ συμμετέχουν στη διαφοροποίηση τη γεωργία και το καθεξή. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι πολιτικοί θύνοντε, οι ερευνητέ, ε, οι ομάδε εκπροσώπηση των γυναικών να λάβουν ενεργό δράση. Γυναίκε στη Γεωργία λοιπόν, Ω προ το θέμα αυτό πρέπει να, να παραδεχθούμε ότι η ανάπτυξη τοπικών ε, αγροτικών αγορών σχετίζονται και με τι περιφερειακέ αγορέ. Και αυτέ οι αγορέ είναι πολύ σημαντικότερε για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μια γεωργικής μετανάλευση και για τι περιοχέ τη υπαίθρου. Ω προ την πρόσβαση στη γη για το ποιοι είναι οι ιδιοκτήτε και ποιοι κάτοχοι ενό αγροτεμαχίου, θα πρέπει να μελετήσουμε τι σημερινέ υπάρχουσε τάσει και να δούμε εάν εξελίσσονται και αν οι εξελίξεις του είναι θετικέ. Όπω προείπα, υπάρχουν κάποια στοιχεία από τι μελέτε που καταδεικνύουν ότι οι γυναίκε μπορεί να έχουν διαφορετικού στόχου εφόσον επλέκονται στη γεωργία λόγω χάρη τη καλλιέργεια που είναι περισσότερο φιλικέ προ το περιβάλλον. Εάν δούμε ότι αυτό ισχύει, θα δούμε ότι μπορεί να συνάδει και με του μελλοντικού στόχου τη ΚΑΠ. Ιδίω στι περιπτώσει όπου οι γυναίκε είναι και κάτοχοι των αγροτεμαχιών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συστηματικότερη στοχοθέτηση των, ε, της κατάρτισης, της στρατηγικής μελέτης και διαχείρισης και των δυνατοτήτων διαχείρισης που έχουν οι γυναίκες σύζυγοι στην Γεωργία προκειμένου να διασφαλίσουμε την συμμετοχή τους στον τομέα που μας ενδιαφέρει. Για την καλύτερη και περισσότερη ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων στη Γεωργία αυτή θα πρέπει να προβλέψουμε και κονδύλια. Δεν είναι απλό όταν οι κυβερνήσεις πρέπει να υποβάλουν προβλέψεις ε, για τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου πριν αποξιολογηθούν και αποτιμηθούν τα προηγούμενα, πριν λήξουν καν. Δεν είναι απλό αυτό, αλλά θα πρέπει οι φορείς υλοποίησης να μελετήσουν τη θέση των γυναικών, να τη λάβουν υπόψη τους, να δουν ποια είναι η συνεισφορά και η συμβολή των γυναικών και πώς τα διδάγματα αυτά μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού. Μπορούμε, απλούστατα κιόλα, να αυξήσουμε την ισορροπία των ε, φύλων όταν δούμε αν υπάρχουν ήδη θετικά αποτελέσματα σε ένα πρόγραμμα. Αυτό τίνει να είναι τάση ούτως ή άλλως σε οργανώσεις γεωργών που τα περισσότερα μέλη είναι γυναίκ, ε, άνδρες. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ζητήσουμε και από άνδρες και από γυναίκες να εκπροσωπούν ε, μια επιτυχημένη οργάνωση, ώστε η γνώση και η πείρα των γυναικών να έρχεται στο προσκήνιο. Τέλος, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά ανεπίσημα στοιχεία και από κυβερνητικού και με κυβερνητικού οργανισμού για τη συμβολή των γυναικών στα προγράμματα ανάπτυξη τη υπαίθρου. Κάποιε συγκριτικέ ποιοτικέ ε, μελέτε με συνεντεύξει ε, των απλών ανθρώπων που εργάζονται στου τομεί αυτού θα μα διευκόλυνε ιδιαίτερα και θα βοηθούσε να θέσουμε αποτελεσματικότερου στόχου για την ΚΑΠ. Θα μας έδινε επίσης περισσότερες πληροφορίες για τις διαφορές και τις δυσκολίες μεταξύ παλαιών και νέων κατώμελών. Εν τέλει, να σας πω απλώς ότι η θέση των γυναικών στη Γεωργία έχει ήδη αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ανά την Ευρώπη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Tack mycket det var er ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτή και είναι και πολύ σημαντικό να σκεφτούμε το θέμα των φύλων ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στον ιδιαίτερο ρόλο της ανάπτυξης της υπαίθρου. Μιλήσατε για τις περιφερειακές τοπικές αγορές. Αυτό βεβαίως και παίζει έναν σημαντικό ρόλο για την απασχόληση των γυναικών στη γεωργία. Είτε γυναίκες οι οποίες είναι παντρεμένες με αγρότες. Με αυτόν τον τρόπο όλη η οικογένεια μπορεί να ζήσει και να εργαστεί στον ίδιο ε, χώρο, στην ίδια γεωργική εκμετάλλευση. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η Μπετίνα Μποκ. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω το τι έκανε η ομάδα εργασίας μας. Θα περιγράψω καταρχήν την κατάσταση των γυναικών στην Ήπεθρο και θα εστιάσω ιδιαίτερα στις γυναίκες στην Ήπαθρο και όχι μόνο στις γυναίκες που εργάζονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μου ζητήθηκε καταρχήν να καθορίσουμε κάποιους δείκτες που να χαρακτηρίσουν την κατάσταση των γυναικών, εισόδημα, παραδείγματο χάρη, εάν παίζουν κάποιο ρόλο στην λήψη αποφάσεων, την ποιότητα ζωής τους, να δούμε τις διαφορές μεταξύ των περιοχών, των κρατών μελών και των κοινωνικών ομάδων και τέλος να δώσουμε κάποιες ε, συστάσεις για την περίοδο μετά το 2013 βασιζόμενοι στις καλύτερες βέλτιστες πρακτικές. Θα ήθελα καταρχήν να εστιάσω λοιπόν την προσοχή μου σε κάποιες σημαντικά συμπεράσματα και να συζητήσουμε το κατά πόσο αυτό είναι χρήσιμο για την θέσπιση πολιτικών. Πρώτα απ' όλα υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά τη γεωργική περιοχή, όσον αφορά τις κοινωνικές ομάδες, να μιλήσουμε επίσης για την περιθωριοποίηση και τέλος τι θα μπορούσαμε να μάθουμε, πώς θα μπορούσαμε να υποφεληθούμε. Καταρχήν η θέση των γυναικών στην Ήπεθρο. Καταρχήν δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι σε γενικές γραμμές οι γυναίκες στην Ήπεθρο έχουν η πιο μειονεκτική θέση. Οι γυναίκες σε γενικές γραμμές έχουν μειονεκτική θέση. Ε, συμμετέχουν στη μισθετή εργασία, η συμμετοχή τους στην λήψη αποφάσεων και η ικανοποίησή τους και η ποιότητα ζωής τους βεβαίως μας δείχνει ότι υπάρχει αν θέλετε διαφορά με την κατάσταση των γυναικών αλλά η ισότητά τους, η ανισότητά τους δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι ζουν στην Ήπεθρο. Οι γυναίκες βεβαίως που ζουν στην Ήπεθρο σίγουρα ζουν σε μια μειονεκτική, ε, βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση. Ε, προσπαθούμε να βρούμε τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι γεγονός. Η αγορά εργασίας στην Ήπεθρο αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες όπως και η αγορά εργασίας γενικότερα. Υπάρχουν προβλήματα επικοινωνίας, υποδομών και σε πολλές περιοχές δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα απόστασης και απομάκρυνσης. Κατά κάποιο τρόπο η ύπεθρος ε, είναι λιγότερο μακριά και είναι λιγότερο απομονωμένη σήμερα. Και εδώ βλέπετε ένα σκίτσο που δείχνει πραγματικά ότι υπάρχουν επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών και της σύγχρονης ζωής. Οι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας δίνουν νέες δυνατότητες που δεν υπήρχαν ακόμα και μια δεκαετία ε, πριν. Με απλά λόγια θέλω να σας πω ότι πολλές περιοχές της υπαίθρου προσφέρουν σήμερα παρόμοιες δυνατότητες και ευκαιρίες στις γυναίκες όπως και οι αστικές περιοχές και όσον αφορά την ε, αγορά εργασίας αλλά και όσον αφορά την επικοινωνία και την κατάρτιση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εμπόδια και περιορισμοί. Είναι όμως παρόμοια προβλήματα, εμπόδια και περιορισμοί που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες παντού ε, σε άλλες περιοχές και βεβαίως τα προβλήματα αυτά είναι προβλήματα που απορρέουν από τον συνδυασμό κυρίως της οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Οι γυναίκες έχουν προβλήματα ελλειπούς κατάρτισης και πραγματικά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται είναι παρόμοιες, επαναλαμβάνουμε, αυτές των αστικών περιοχών. Όμως, δεν νομίζω ότι μπορούμε εδώ να είμαστε υπεραισιόδοξοι, γιατί υπάρχουν ε, διαφορές και μειονεκτήματα που δεν είναι διαφορές και μειονεκτήματα που οφείλονται στην Ήπεθρο. Υπάρχουν περιοχές ε, παρόλα αυτά στην Ήπεθρο που παραμένουν πολύ απομακρυσμένες και πολύ απομονωμένες. Η απομόνωση αυτή μπορεί να οφείλεται και σε κοινωνικούς παράγοντες οι περιοχές αυτές, οι οποίες κυρίως εξαρτώνται για την ανάπτυξή τους από την γεωργία, με πολλές θέσεις απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και όχι στον τομέα των υπηρεσιών, με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και με προβλήματα ποιότητας ζωής. Αν θέλετε, αυτή η απομάκρυνση δεν είναι καθαρά γεωγραφική απομάκρυνση, δεν είναι μια απομάκρυνση και απομόνωση που οφείλεται στην απόσταση, αλλά σε όλους αυτούς τους παράγοντες. Άρα, όταν μιλάμε για ύπεθρο, δεν εννοούμε καθαρά ύπεθρο. Η απομάκρυνση και η απομόνωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση. Υπάρχουν ε, περιοχές της ύπεθρου, οι οποίες είναι εύκολες στην πρόσφαση και βρίσκονται πολύ κοντά σε αστικές περιοχές. Οι περισσότερες βρίσκονται στο βορρά και στην δυτική Ευρώπη. Και αυτές που είναι πιο περιφαριακές και απομονωμένες είναι στη νότια ανατολικη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί αντιμετωπίζονται και οι μεγαλύτερες δυσκολίες. Αυτό που θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω είναι ότι η μειονεκτική θέση αυτών των ε, περιοχών αν θέλετε ε, μας οδηγεί στο θέμα της ε, περιθωριοποίησης. Λίγες δυνατότητες μεταφορών, λίγες δυνατότητες πρόσβασης και στους πελάτες και στις αγορές. Πρόκειται επίσης για περιοχές με κακή επικοινωνία, κακή πρόσβαση ή ελλειπή πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες, στα δίκτυα, αλλά και με πολύ λιγότερη κοινωνική ζωή. Τα άτομα που ζουν στις περιοχές αυτές είναι λιγότερο συνηθισμένοι στις ε, κοινωνικές ε, σχέσεις, στην κοινωνική ανάπτυξη, είναι λιγότερο αισιόδοξοι και δεν έχουν εμπιστοσύνη στην σύγχρονη ζωή. Εν πάση περιπτώσει δεν πιστεύουν ότι θα μπορέσουν εύκολα να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την σύγχρονη ζωή. Σε αυτές τις περιοχές ε, παρατηρούμε και πολύ πιο έντονα φαινόμενα ανισότητας μεταξύ των φύλων με λιγότερη απασχόληση, λιγότερες υπηρεσίες και κοινωνική απομόνωση. Επιπλέον σε αυτές τις περιοχές ε, με συσσωρευτικό τρόπο προστίθενται και προβλήματα υποανάπτυξης της Υπήρου, της Υπέθρου. Βλέπουμε την ίδια ώρα ότι η χαμηλή ποιότητα ζωής, η έλλειψη αισιοδοξία, στήριξης είναι ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει όχι μόνο τις γυναίκες αλλά και τους άντρες και κυρίως τους νέους. Ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες όλων αυτών για την κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013. Καταρχήν, όταν παρατηρείται αυτή η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αυτό παρατηρείται κυρίως σε περιοχές με υποανάπτυξη και κοινωνικά προβλήματα στην ύπαρχο. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα περιθωριοποίησης, αλλιώς οι γυναίκες θα συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές, ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή. Αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν το κάνουν απλώς οι γυναίκες, αλλά και οι άνδρες και οι νέοι. Αυτό ενδυναμώνει τα προβλήματα στις ίδιες αυτές περιοχές οδηγώντας πολλούς νέους επιχειρηματίες και νέους ε, γεωργούς στο να τις εγκαταλείψουν. Θα πρέπει λοιπόν καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να διδοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις ε, περιοχές, τις απομακρυσμένες. Υπάρχουν προβλήματα ανισότητας φύλων, όχι μόνο βεβαίως στη... Και η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές τις περιθωριακές, περιφερειακές περιοχές ενισχύοντας την κινητικότητα, επενδύοντας στα δίκτυα, στην ποιότητα ζωής, κάνοντας τις περιοχές αυτές ελκυστικές για τις γυναίκες και για τους νέους, έτσι ώστε να παραμείνουν εκεί, να δεσμευθούν, να επενδύσουν και να μην θέλουν να τις εγκαταλείψουν. Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις αυτές πριν ε, περιμένουμε από όλους αυτούς τους ε, άνδρες και γυναίκες να δεσμευθούν και να παραμείνουν. Όταν μιλάμε για ισότητα των φύλων, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες πρόσφατες εμπειρίες κοινών ε, προγραμμάτων ανάπτυξης της υπέρτου και θα ήθελα πραγματικά να πω ότι για προγράμματα που μας έδειξαν τρομερές ελλείψεις και αδυναμίες. Τα αποτελέσματα είναι κοινά. Υπάρχουν ελάχιστα προγράμματα που απευθύνονται στις γυναίκες και κυρίως αυτά προστίθενται στην γενικότερη προσπάθεια ανάπτυξης της υπαίθρου. Ποτέ δεν είναι εξειδικευμένα προγράμματα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα πρέπει και με γεωγραφικό και εδαφικό τρόπο να αντιμετωπιστεί το θέμα της ισότητας των φύλων. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι ειδικέ ανάγκες της κάθε περιοχής. Κατόπιν να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές να ενισχυθούν οι οργανώσεις των γυναικών πέρα από τα περιφερειακά αυτά σύνορα και δομές, να δημιουργήσουμε δίκτυα ασφαλείας, παραδείγματο χάρη για θέματα ασφάλειας, βίας κατά των γυναικών και οι οργανώσεις ε, των γυναικών μπορεί εδώ να παίξουν και ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά την συμμετοχή των μελών τους σε αυτά τα περιφερειακά προγράμματα. Πολλές φορές βλέπουμε ότι η εκπροσώπηση ε, των γυναικών ε, είναι ελλειπής σε πολλά τέτοια προγράμματα ανάπτυξης. Θα ήταν πολύ σημαντικό οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές να ε, είναι αρμόδιες να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι κάπου γίνεται ένας απολογισμός αυτών των ε, αποτελεσμάτων και να υπάρξει και μια συντονιστική αρχή τι πετύχαμε και τι ακόμα πρέπει να κάνουμε. Γιατί σήμερα έχουμε ελάχιστο, ε, ελάχιστη δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων όλων αυτών των προγραμμάτων. Τελειώνοντας, θα σας αναφέρω μία από τις αγαπημένες μου ενασχολήσεις, που είναι η συλλογή στοιχείων, στατιστικών στοιχείων και η έρευνα. Έχουμε πολλά στοιχεία για πολλούς τομείς, ενώ πραγματικά για τον τομέα που μας αφορά εδώ η πληροφόρηση είναι εξαιρετικά λίγη. Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που να αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες. Αυτό μας ε, εμποδίζει να βασιστούμε σε συγκρίσιμα στοιχεία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα. Πολλές ε, ερωτήσεις λοιπόν παραμένουν εκκρεμείς, παραμένουν ανοιχτές. Η ταυτότητα των ε, γυναικών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, την Ήπεθρο, η μετανάστευση. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε στοιχεία που να αφορούν τις μετακινήσεις γυναικών αλλά και ανδρών μεταξύ των περιφερειών. Δεν ξέρουμε πόσες εγκαταλείπουν την Ήπεθρο ή πόσες επιστρέφουν ή αποφασίζουν να εγκατασταθούν στην Ήπεθρο. Όλες αυτές λοιπόν οι πολύ σημαντικές ερωτήσεις δεν έχουν απαντηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά. μας επιβεβαιώνουν ότι χαρακτηριζόμαστε από άγνοια σε πολλά σημεία. Για παράδειγμα, ε, ε μάλλον και πρέπει να απαντήσουμε ε, σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Κυρία Γέγκλε έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις δύο εξαιρετικά σημαντικές παρουσιάσεις οι οποίες μας οδηγούν ε, σε περαιτέρω σκέψη, σε νέα ερωτηματικά. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει μία σειρά σημαντικών αποφάσεων όσον αφορά την ίση αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών τις ίσες ευκαιρίες. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα. Για μένα, αλλά νομίζω για την Επιτροπή μας, όταν επεξεργαστήκαμε την έκθεση που αφορά το θέμα αυτό, εξετάσαμε μία σειρά ερωτημάτων. Καταρχήν, Η Ισπανική Προεδρία είχε θέσει τον ρόλο των γυναικών ε, στον αγροτικό τομέα σαν μία από τις τρεις προτεραιότητές της. Δεν θέλω να εγκαταλειφθεί το θέμα αυτό και στη συζήτηση που είχαμε με τον Επίτροπο πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας για τον ρόλο των γυναικών είχε σαν κύριο θέμα την κοινή αγροτική πολιτική και το θέμα των γυναικών και δεν μιλάω τώρα μόνο για τις γυναίκες που είναι στον τομέα της γεωργίας αλλά όλες τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο είναι εξαιρετικά σημαντικός αλλά και από πολιτικής απόψεως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι συνθήκες οι οποίες τους επιτρέπουν να παραμείνουν στην Ήπεθρο, να συνεργαστούν για την ανάπτυξη αυτής της Ήπεθρου και είμαστε σήμερα και σε θέση να εξετάσουμε αυτήν την ποιότητα ζωής, να δούμε τι δυνατότητες χρηματοδότησης μπορούμε να τους προσφέρουμε. Εσείς είπατε ότι πρόκειται για το δεύτερο πυλώνα, ότι υπάρχει η επικουρικότητα, ότι τελείως διαφορετικά αντιμετωπίζουν το θέμα τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. Παρόλα αυτά, μέχρι το 2013 ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, μετά όμως δεν πρέπει να χαθεί η δυνατότητα που έχουμε σήμερα. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό μετά το 2013 γιατί πέρα από την κατάσταση της ιδιοκτησίας ή της άμεσης εκμετάλλευσης διαχείρισης, Πιστεύω θα πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα θέματα αυτά που άπτονται του δεύτερου πυλώνα. Το θέμα της συγκέντρωσης. Εγώ είμαι από το κρατήδιο της Βάδης Βουτεμβέργης και διαπιστώνω καθημερινά ότι διαρκώς οι προτάσεις που έρχονται από τις αστικές περιοχές είναι πάντα πολύ πιο έντονες και πολύ πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές θα έλεγα. Αγνοούμε συστηματικά τα προβλήματα των ε, γεωργικών περιοχών της Υπέθρου. Και αυτό φαίνεται και στη χρηματοδότηση και ιδιαίτερα ο ρόλος των γυναικών είναι κάτι που θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο αυτών που μας απασχολούν. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στην κοινωνία, στην οικονομία θα πρέπει να υπογραμμιστούν. Η έκθεση που προετοιμάζουμε σαφώς θα πρέπει να συμπεριλάβει όλες αυτές τις πτυχές. Πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας. Όμως, πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας η οποία συμπεριλαμβάνεται στην γενικότερη δραστηριότητα εισηγήσεων και εκθέσεών μας. Και οι προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της υπαίθρου θέλω να είναι μια δραστηριότητα η οποία να έχει στο επίκεντρό της ε, τις γυναίκες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε πώς εκπροσωπούνται οι γυναίκες στις επαγγελματικές οργανώσεις. Πολύ σπάνια τις βλέπουμε στο προσκήνιο. Εμείς μέχρι το τέλος Μαρτίου θα επεξεργαζόμαστε την έκθεση αυτή και ο κύριος στόχος μου είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση στις ε, οργανώσεις, τις αντιπροσωπευτικές των γυναικών της υπαίθρου μία συζήτηση η οποία πραγματικά θα ενισχύσει τις προτάσεις των γυναικών. Πιστεύω ότι οι γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις είναι σε θέση να μας υποβάλουν προτάσεις και μετά τη Λισαβόνα έχουμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε αυτές τις ε, προτάσεις που θα προκύψουν. Σας καλώ λοιπόν όλους να κινητοποιήσετε αυτές τις ε, οργανώσεις. Ζητώ από όλους τους συναδέλφους εδώ να εμπλουτίσουν την συζήτηση και την έκθεση αυτή. Και σας το λέω με μεγάλη σαφήνεια. Θα ακολουθήσουμε την ομαλή μας διαδικασία εργασίας, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πιστεύω ότι με την έκθεση αυτή στρέφουμε τον προβολέα στις γυναίκες αυτές που ζουν και εργάζονται στην Ήπεθρο και στον τομέα της γεωργίας. Ευχαριστούμε κυρία Γέγκλερ. ο λόγο στην κυρία Ταντζίλα. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος τα ονόματά σας, αλλά προσπαθώ. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω για όλες αυτές τις παρουσιάσει γιατί πραγματικά ε, καταδεικνύουν το ρόλο της γυναίκας ε, στην γεωργία. Είναι ένας τομέας ο οποίος δίνει ευκαιρίες παρόμοιες με αυτές που δίνει μια πόλη σε μια γυναίκα και ταυτόχρονα η γεωργία τους επιτρέπει να βοηθούν την οικογένειά τους οικονομικά πολύ αποτελεσματικά. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για, την, για τις γυναίκες είτε χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους είτε ε, χρησιμοποιούν ε, μεθόδους πιο παραδοσιακές ε, που απλώς επιτρέπουν, τους επιτρέπουν να επιβιώσουν. Ε, θα μπορούσα να σας δώσω κάποιες ιδέες, κυρία Γέγκλε, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη της Επιτροπής μας στην Ρουμανία. Στο πρόγραμμα είχαμε μια επίσκεψη σε μια παραδοσιακή, μικρή παραδοσιακή εκμετάλλευση σε μια ορεινή περιοχή. Και εκεί οι ευρωβουλευτές είδαν ποιε είναι οι δυσκολίες που, αντιμετωπίζουν, που αντιμετωπίζει μια μικρή οικογένεια με γονεί και τρία παιδιά. Ε, και η Μπετ Κέγλε θέλησε να τους ευχαριστήσει για την ε, ε, φιλοξενία τους και αντιλήφθηκε ότι η σύζυγος είχε εγκαταλείψει την παρέα. Ο σύζυγός της της είπε ότι ε, η γυναίκα του χρειάστηκε να πάει να φροντίσει τα, λόγια που, τα ζώα που είχαν γυρίσει από ε, τη βοσκή τους. Και η κυρία Γέγκλε τον ρώτησε έτσι είναι πάντοτε οι γυναίκες ε, δουλεύουν και οι άντρες δρέπουν τις δάφνες είμαι σίγουρη ότι η κυρία Γέγκλη θα δώσει έμφαση στις γυναίκες γιατί ε, οι γυναίκες ε, χρειάζονται και αυτές δάφνες όπως και οι άντρες. Ελπίζω ότι θα τις μεταχειριστούμε τον ίδιο τρόπο. Η δυσκολίες των γυναικών ε, είναι κοινέ για όλη την Ευρώπη. Και ε, τα προβλήματα των γυναικών είναι παρόμοια με αυτά των ανδρών. Θα πρέπει να τα, πολλά από αυτά να τα αντιμετωπίσουμε με κοινό τρόπο. Και χρειαζόμαστε έναν προϋπολογισμό επαρκή. Χρειαζόμαστε καινούρια μέσα τα οποία θα προωθήσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και στην υπεθρο. Ευχαριστώ. Nästa talare är herr Ευχαριστούμε κύριο Σταραμπέλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. vous ai exposé euh, très éloquent. Il a moins de bourdonnement, je crois, ici. Ήταν ιδιαίτερα ευλάδης οι ε, ομιλητρίε μα, παρόλο που ήταν σύντομε, για την πρώτη παρουσίαση που επικεντρώθηκε στο ρόλο των γυναικών στη Γεωργία με αριθμού όπω 41% του εργατικού δυναμικού. Ε, ναι, ε, είναι δεν είναι ακριβώ μειοψηφία, είναι σχεδόν ισότιμη η προσώπηση Όμω, όπω επιβεβαιώσατε, το 38% έχουν ε, το καθεστώς συζύγων ε, βοηθητικού προσωπικού. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρέπει να δοθεί αγώνας στο μέλλον για μεγαλύτερη, για περισσότερα και ίσα δικαιώματα και σε ό,τι αφορά τα κοινά δικαιώματα στην ιδιοκτησία, του τίτλου ιδιοκτησία, εδώ θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κατά πόσον ε, η δύναμη των γυναικών οδεύει στην, ε, στις ζωικές δραστηριότητες αυτές καθεαυτές. Εάν υπάρχουν δύο εκμεταλλεύσεις με ίδια δραστηριότητα και τα ίδια έσοδα, δεν έχει σημασία ποιος έχει την ιδιοκτησία. Όμως την ημέρα που δεν θα ισχύει αυτό πια, η γυναίκα θα βρίσκεται σε προσωρινή κατάσταση επισφάλεια, εκτό αν έχει δικαίωμα στο τρίλο ιδιοκτησία. Τότε θα εξασφαλίσει τα δικαιώματά τη και θα είναι προστατευμένη. Κάτι που δεν ισχύει σήμερα. Έπειτα, πραγματικά να υπάρξει αναγνώριση της κατηγορίας γυναίκας Γεωργού ως ε, ιδιοκτήτριας και ανεξάρτητης εργαζομένης και για να έχει και συνταξιδοτικά δικαιώματα στη χώρα μου, το Βέλγιο, που έχει ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας ε, που κάποιοι το θεωρούν υποδειγματικό, με πολλά ελαττώματα αλλά πολλά σίγουρα, με πολλά μάλλον αρνητικά αλλά και πολλά θετικά. Ξέρουμε ότι η γυναίκα όταν ε, πρέπει να πάρει σύνταξη από το γεωργικό τομέα παίρνει ελάχιστα δεν μετράνε οι ώρες εργασίας της ως συνταξιδοτικά δικαιώματα, ούτε σε πρώτερη συνταξιοδότηση, ούτε ως, στη σύνταξή της τελικά. Και έχουμε προσπαθήσει πολύ στο Βέλγιο σε αυτό το τομέα, έχουμε επιτελέσει κάποιους πρόοδους, αλλά και άλλα πρέπει να γίνουν. Και το τρίτο που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι και συνάδελφος πολύ καλά τα είπε, κυρία Νταντσίλα, ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε τις προκαταλήψεις. Οι άντρες οδηγούν τα τρακτέρ και οι γυναίκες αρμέχουν τις αγελάδες. Αυτό δεν ισχύει πια. Μπορεί εγώ οδηγούσα μια Ferguson 136. Δεν υπάρχουν αυτά πια με ε, θερμάστρα και καυστήρα και με αναγκαστική χρήση γυαλιών και προστατευτικά για τα αυτιά. Δεν υπάρχουν τέτοια τρακτέρ, μπορούν να το οδηγήσουν και γυναίκε. Και προκαταλήψει αυτέ αυτές υφίστανται. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε τι υπάρχουσες τάσει. Και θα πρέπει οι γεωργικέ εργασίε που αυτή τη στιγμή είναι μονοπόλιο των ανδρών να μοιράζονται με τρόπο ισότιμο μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τώρα, για την παρουσίαση που αφορούσε τι γυναίκε και την παρουσία του στι περιοχέ τη Υπέθρου. Υπάρχουν διαφορετικέ περιοχέ στην Υπέθρο, σαφώ. Δεν είναι μία Υπέθρο. Υπάρχουν κάποιε περιοχέ που είναι περισσότερο ευνοούμενε, στα προάστια των πόλεων, όχι μακριά από τι πόλει τέλο πάντων. Υπάρχει καλό δικό δίκτυο. Όμω, οι περιοχέ αυτέ θα μπορούσαν να ονομάζονται γεωργαστικέ ή αστικογεωργικέ. Είναι ίσω περισσότερο ελκυστικέ και κατοικούνται από όσου ε, λόγω των αστικών πιέσεων εγκαταλείπουν την πόλη και πάνε να ζήσουν στην εξοχή. Όμω, ε, εδώ η διαφορά δεν φαίνεται να είναι διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά κοινωνική ε, ανακατανομή. Διότι στι περιοχέ αυτέ, μαζί με την πίεση των τιμών των κατοικιών, είτε μιλάμε για ενοικίαση είτε για ιδιοκτησία και επειδή έχουμε άκρα το, άκρατη απελευθέρωση και φιλελευθερισμό και στις δημόσιες υπηρεσίες. Λιγότερες ταχυδρομικές, σιδηροδρομικές ε, υπηρεσίες, λιγότερα λεωφορεία. Εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά, διότι όταν έχουμε μια οικογένεια με δύο γονείς, χρειάζεται οπωσδήποτε και ένα αυτοκίνητο, ένα όχημα, δύο μάλλον οχήματα για να ζει κανείς στην εξοχή. Πόσο επισφαλή λοιπόν η θέση τη γυναίκα στην Ήπεθρο, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, όταν υπάρχει ένα διαζύγιο. Η γυναίκα αναλαμβάνει την κυδαιμονία των παιδιών. Οι γονεί χωρίζουν λοιπόν, τα εισοδήματα μοιράζονται στη μέση. Όσα κερδίζει ο ένα ε, υπολογίζεται ότι κερδίζει και ο άλλο, όμω είναι πολύ διαφορετικέ οι δαπάνε. Και το αυτοκίνητο που πληρώνει, η γυναίκα και τα έξοδα για τη στέγαση. Οι γυναίκε λοιπόν είναι περισσότερο θύματα διότι έχουν ακριβώ και την ε, κυδαιμονία, το βάρο των παιδιών. Πρέπει να κάνουν περισσότερε μετακινήσει. Ακόμη και αν έχουν ε, κάπου να μείνουν, πρέπει να αναλάβουν το βάρος αυτό, εκτός και αν νοικιάσουν. Και βεβαίως υπάρχουν και χώρες με λιγότερο αναπτυγμένο οδικό δίκτυο, με περιοχές της υπαίθρου που είναι πραγματική υπαίθρος. Ε, εκεί Υπάρχει το θέμα της ε, μαζικής αποχώρησης από την έξοδο. Αλλά εκεί υπάρχουν, από την Ήπεθρο, συγγνώμη, εκεί υπάρχουν όμως διαφορετικά προβλήματα. Οπότε ίσως υπάρχει και, και περιθώριο μελέτης. Βεβαίως είναι θέμα και ισότητας φύλων, αλλά είναι κυρίως θέμα κοινωνικής ανάμειξης. Εγώ νομίζω ότι αυτό αφορά περισσότερο τις περιοχές της Πέθρου κοντά στις πόλεις και αυτούς που έχουν λιγότερα μέσα οικονομικά. Για να μην φτάσω στα προάστια. Θα πρέπει λοιπόν να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε θα το γυρίσω στα αγγλικά, ζητώ συγγνώμη, αλλά όταν μιλάω ουγγρικά οι ερωτήσεις μου είναι τόσο αστείες φαίνεται που κάνουν ακόμα και τον Επίτροπο να γελάει. Οπότε ας μιλήσω αγγλικά. Μιλούμε για τις γυναίκες στις εκμεταλλεύσεις, μικρές εκμεταλλεύσεις πολύ συχνά Δεν νομίζω ότι ε, στις ε, οικογενειακέ εκμετάλλευσει υπάρχει σημαντική, σημαντικό πρόβλημα ανισότητας των φύλων. Το πρόβλημα είναι πιο πολύ στις βιομηχανικέ εκμεταλλεύσεις, δηλαδή στη σύγχρονη γεωργία ε, που παράγει πρώτε ύλε για τη βιομηχανία. Σε αυτού του τύπου τη εκμεταλλευση, πολύ σπάνια βρίσκουμε γυναίκε. Και θα ήθελα να μα δώσετε μερικά στοιχεία γι' αυτό. Από όσο γνωρίζω τις στατιστικές, αλλά και η δική μου προσωπική εμπειρία είναι προς αυτή την κατεύθυνση ότι σε αυτού του τύπου της εκμεταλλεύσης ε, η απασχόληση των γυναικών είναι σχεδόν μηδενική. Έχω δίκιο ή όχι. Και θα ήταν σωστό ασφαλές συμπέρασμα ότι χάνοντας οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ε, οι γυναίκες χάνουν σε ευκαιρίες απασχόλησης, ότι δηλαδή η μετάβαση από την ε, ε, οικογενειακή γεωργία στη βιομηχανική γεωργία θέτει σε κίνδυνο την απασχόληση των γυναικών, είναι σωστό συμπέρασμα αυτό. Άλλη παρατήρηση αυτή τη φορά είναι το ότι είπατε πως υπάρχουν πολύ λίγα ποσοτικά στατιστικά στοιχεία για τις γυναίκες στις ε, γεωργικές περιοχές, σε αγροτικές περιοχές ή στη γεωργία. Θα ήθελα να προτείνω και σε εσάς και στην κυρία Γέγκλε που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα, τις απόψεις των μελών. Ο, να πω λέω ότι οι έρευνες ε, για την... Ε, ε, ότι μπορείτε να ρωτήσετε τις ίδιες τις γυναίκες και να κάνετε ποιοτικέ έρευνες. Ελάτε στην Ουγγαρία, ελάτε στην Ανατολική Ουγγαρία, θα σας βοηθήσω να, να ρωτήσουμε μαζί ε, τις γυναίκες για τη βία, για το φόβο που μπορεί να έχουν, που να τους προκαλεί η βία για την έλλειψη των μέσων μαζικής μεταφόρας. Μπορείτε να τις ρωτήσετε και νομίζω ότι είναι κομμάτι του έργου μας. Γιατί πράγματι δεν έχει γίνει πολλή έρευνα και η κατανόηση του ρόλου των γυναικών στις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρουμανία, Ουγγαρία κλπ. Ε, είναι πολύ ελλειπής. Γιατί τα συμπεράσματα από τη Γερμανία ή τη Βρετανία ή άλλες χώρες της Δυτική Ευρώπης δεν εφαρμόζονται άμεσα στην Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. And first of all, thank you to the two ladies who made... Ευχαριστώ πολύ για τις δύο παρατηρήσεις Σίγουρα δεν έχουμε πολλές ε, πληροφορίες και αυτές που έχουμε πολύ συχνά δεν είναι κατανεμημένες σαν αφήλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσα είπατε μας δίνουν τροφή για σκέψη. Ένα από τα κρίσιμα σημεία ε, τα οποία θίξατε είναι η άμεση σύνδεση της οικογένειας με την εκμετάλλευση. Πάντοτε μιλούμε εδώ και αλλού για το μοντέλο της ευρωπαϊκής οικογενειακής ε, ε, Εκμετάλλευση. Και η ερώτηση είναι πώ η κοινή αγροτική πολιτική συνεισφέρει σε αυτό. Ο George ε, που ε, συνέταξε την πρώτη μας έκθεση για την ΚΑΠ μετά το 2013. Ε, αν τη διαβάσουμε αυτή την έκθεση δεν θα δούμε τίποτα για τις γυναίκες. Δεν θέλω να τον κατηγορήσω. Ναι, με κατηγορείς, της λέει ο κ. Λάιον. Όχι, δεν σε κατηγορώ. Ε, γιατί δεν είχαμε δώσει έμφαση σε αυτό το θέμα ως τώρα. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα το κάνουμε. Πολύ συχνά ε, τις βάζουμε στο περιθώριο τις γυναίκες και δεν αναγνωρίζουμε το έργο τους όταν χαράσουμε πολιτική. Μιλήσατε επίσης για την ένταξη του φίλου στις υπόλοιπες πολιτικές και σίγουρα ε, αυτό το mainstreaming είναι ελλειπές προς το παρόν. <clears throat> Υπάρχει και η ερώτηση γιατί να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στη Γεωργία. Ε, αυτό θεωρούμε ότι είναι θετικό και πράγματι θα πρέπει να το κάνουμε θετικό, αλλά χρειάζεται να απαντήσουμε γιατί πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στη Γεωργία. Ε, είναι σαν να ρωτάμε βέβαια γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική. Εμένα στη χώρα μου το 13% των ε, βουλευτών μας είναι γυναίκες μόνο. Οπότε μα ρωτάνε πολύ συχνά γιατί χρειάζομαστε περισσότερε γυναίκε, παίρνουν καλύτερε αποφάσει οι γυναίκε. Εγώ του απαντάω όχι. Πολύ συχνά όμω παίρνουν διαφορετικέ αποφάσει. Χρειαζόμαστε μια ισορροπία στην λήψη αποφάσεων. Το ίδιο ενδεχομένω χρειαζόμαστε και στι πρακτικέ, στι γεωργικέ πρακτικέ που ασχολούνται. Αυτό ίσω θα μα βοηθούσε να ισορροπήσουμε και όλο τον τομέα της γεωργίας. Και βέβαια γιατί θέλουμε ισότητα και καλύτερη ε, και, βέβαια η τελική απάντηση είναι θέλουμε περισσότερες γυναίκες γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη ισότητα και περισσότερη πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση. Μετά το θέμα της ε, ε, τοπικής προσέγγισης ε, στην ισότητα των γυναικών. Ε, το πρόβλημα δεν είναι το πού βρίσκονται οι γυναίκε, ε, δηλαδή αν βρίσκονται σε περισσότερο ή λιγότερο υγειοικές ή απομακρυσμένες πολιτικές, αλλά στην απομόνωσή τους. Γιατί πολύ συχνά στι περιοχές όπου βρίσκονται δεν υπάρχουν βασικέ δημόσιες υπηρεσίε, αγαθά κλπ. Το θέμα σχετίζεται επίση με την εδαφική συνοχή και το φύλλο θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτή την πολιτική. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πτυχή φύλου στην εδαφική συνοχή. Θα πρέπει να το δούμε πολύ κοντά, το είπε η κυρία Γέγκλε και πιστεύω ότι μέσω της έκθεσης θα μπορούσαμε να το τονίσουμε. Συμφωνώ επίσης και με ορισμένου άλλους που είπαν ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με τις γυναίκες αγρότησες, με τις οργανώσεις τους για να μάθουμε από την εμπειρία τους. Πολύ συχνά συντάσσουμε κανονισμούς, αλλά ο λαός είναι αυτός ο οποίος ζει με τους κανονισμούς. Θα πρέπει να μιλήσουμε με τις αγρότησες. Είναι πολύ επίκαιρη συζήτηση αυτή, γιατί είμαστε κοντά στην αναθεώρηση της ΚΑΠ. Είναι σημαντικό όμως το θέμα των γυναικών να μην μπει σε ένα κουτί απομονωμένο μόνο του, ε, και γιατί μετά θα περιθωριοποιηθεί. Θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα της ε, μεγαλύτερης πιο πλατιάς εικόνας. Ο Μάρκ Ταραμπελά μίλησε για την αξία του έργου των γυναικών. Παραδοσιακά, στο παρελθόν, η το έργο των γυναικών ήταν αφανές και σχολιάστηκε το θέμα των συντάξεων των αγροτησών. Ε, είχα καλέσει μία, ε, σε μία ακρόαση και ε, μου τόνισε το πόσο, πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες να έχουν τη δική τους σύνταξη όταν μεγαλώσουν που να μην εξαρτάται από τη σύνταξη του άντρα τους. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να περιθωριοποιήσουμε το θέμα, θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής μας για την, όταν συζητάμε την αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2013. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Λόγου χάρη, γιατί χρειαζόμαστε τις γυναίκες στη Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακριβώς θέλουμε να παραμένει ζωντανή η γεωργία. Χρειαζόμαστε και άντρες και γυναίκες στη γεωργία. Ιδάλλως, μια γενιά αργότερα δεν θα υπάρχει γεωργία αν δεν υπάρχουν γυναίκες σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Πριν αρχίσουμε να γινόμαστε αρνητικοί για το ρόλο των γυναικών στη Γεωργία. Να θυμίσω ότι γίνεται στην Βόρεια Ιρλανδία από όπου προέρχομαι. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε υπουργό υπεύθυνο για την Γεωργία που είναι η γυναίκα. Και υπάρχει και υπουργό στη Βόρεια Ιρλανδία. Ω Ευρωβουλευτή έχω ασχοληθεί εκτεταμένα με τα θέματα ενέργεια και γεωργίας και αναγνωρίζω πολύ καλά τη φωτογραφία από την αγορά που δείξατε, το φόρουμ. Και έχω και ένα αντίτυπο της ε, εφημερίδας αυτής των Γεωργών της Βόρειας Ιρλανδίας, της οποίας εκδότρια είναι γυναίκα. Ας μην γινόμαστε λοιπόν αρνητικοί. Υπάρχουν κάποια πολύ καλά παραδείγματα για το πώς οι γυναίκες γίνονται υποδείγματα και παραδείγματα προς μίμηση και εργάζονται και σε αυτόν τον τομέα όπως και σε άλλους σε έναν ανδροκρατούμενο εντός εισαγωγικών κόσμο. Απλώς θέλω να επικεντρωθώ στα εξής. Εγώ μεγάλωσα σε ένα μικρό αγρόκτημα στη Βόρεια Ιρλανδία. Ήταν μια εκμετάλλευση που απασχολεί σε μερικό χρόνο. Ο πατέρας μου έφευγε για να δουλέψει τη μέρα και η μητέρα μου όταν εκείνο έλειπε έκανε τι γεωργικές εργασίες και αυτό ήταν ο ρόλος πολλών γυναικών εκείνη την ε, εποχή. Και ακόμη είναι. Όμως εκείνη είχε ένα βασικό στόχο για τα τρία παιδιά της και αυτό ήταν να μορφωθούν για να μην κάνουν ό,τι ζούσε η ίδια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την όλη κατάσταση τη ε, Γεωργία στη Βορειοελλανδία, την εποχή που εγώ μεγάλωνα. Η κατάσταση δεν ξέρω αν έχει αλλάξει παντού. Πάντω, η, η εποχή όπου οι γυναίκε στην Ήπεθρο είναι καλύτερα μορφωμένε, έχουν περισσότερη κοινωνική κινητικότητα και μπορούν να δουλέψουν εκτό εκμετάλλευση από επιλογή τη ζωή του, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα μιλήσαμε για τις γυναίκες στην Ήπεθρο. Κατά τύχη απόψε θα συμφάγω με εκπροσώπους μιας ένωσης από τη Βόρεια Ελλανδία που εκπροσωπούν ένα δίκτυο γυναικών και οι οποίοι χρησιμοποιούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα διευθυντικά ταμεία που τους έρχονται από την υπηρεσία για την κατάρτιση και την εκπαίδευση προκειμένου να βελτιώσουν την κατάρτιση και την πρόσβαση στην κατάρτιση για τις γυναίκες της Ήπεθρου. Αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό και χρηματοδοτείται από τα διευθυντικά ταμεία. Τον ερχόμενο μήνα, τον Οκτώβριο, Έχω μια ομάδα στήριξης ε, μάλλον θα έρθει μια ομάδα στήριξη ε, γυναικών της Υπέθρου στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί μου. Ας έρθει να τη συναντήσει κυρία Γέκλε, γιατί είναι ένας πολύ ζωντανός, εύρωστος οργανισμό τη Βορείου Ιρλανδίας. Ξέρω ότι ίσως δεν το έχετε ξανακούσει τον οργανισμό αυτό, αλλά θα μείνουμε σε επαφή. Είναι σημαντικότατο. Οι γυναίκες αυτές ανέλαβαν ε, την πρωτοβουλία να έρθουν στο Ευρωκοινοβούλιο για να δουν τι γίνεται και από εδώ. Να μην υποτιμούμε λοιπόν τον ε, ρόλο των ε, γυναικείων οργανώσεων όπως αυτές και για την συνομιλία τους με τους κοινωνικούς εταίρους και για την κοινωνική κινητικότητα και για την δημιουργία εισοδήματος σε έναν ανδροκρατούμενο τομέα και για την απασχόληση. Υπάρχουν, ακούσαμε ανεπίσημα στοιχεία, για γυναίκες που απασχολούνται απευθεία στον τομέα της γεωργίας και κάποια δεδομένα δείχνουν ότι ιδίω στην κτηνοτροφία έχουν ε, λαμπρό ρόλο οι γυναίκες στις διάφορες τοπικές κοινότητες. Ολοκληρώνοντας, ένα από τα τελευταία, τελευταία σχόλια που ακούσαμε ήταν για τις περιοχές και τις προσδοκίες μας για τις γυναίκες. Να στηρίξουμε την κινητικότητα, να επενδύσουμε στην ποιότητα της διαβίωσης, να επενδύσουμε τους γεωργούς ότι αρκεί να μείνουν στις περιοχές τους και να επενδύσουν. Αυτό δεν διαφέρει ούτε για γυναίκες ούτε για άντρε. Στη Βορειολανδία είχαμε ένα πολύ θλιβερό ιστορικό αυτοκτονιών από τον πληθυσμό της υπαίθρου και λόγω των πιέσεων που ζουν από την διαχείριση επιχειρήσεων στον τομέα αυτό και σε τόσο δυσχερείς συνθήκες. Οικονομικές δηλαδή συνθήκες. Είναι δύσκολο τους νεαρούς άντρες να τους πείσουμε ότι μπορούν να ζήσουν καλά στην Ήπεθρο, να πετύχουν επιχειρηματικά και να έχουν και δουλειά. Και αυτό λοιπόν να μην το ξεχνάμε. Και ένα τελευταίο ακόμη ζήτημα. Μιλήσαμε για τα ζητήματα ιδιοκτησία και ούτω καθεξής. Για τη γη. Νομίζω ότι πραγματικά κινδυνεύουμε να περάσουμε σε περιορισμό της εθνική αρμοδιότητας και να ισοπεδώσουμε τις πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Τελευταίο τελευταίο σχόλιο. Δεν θέλω τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου που έμπλεξαν τη Βόρεια Ιρλανδία σε ε, πολλά διοικητικά τερτύπια να αυξηθούν ε, και να επιβαρυνθούν και άλλο. Να μην γίνουν ένα δυσχερές μέσο, δυσκίνητο, προκειμένου να ωφεληθεί η ισότητα των φίλων. οι μελέτες και οι έρευνες ας μην πολλαπλασιάζονται για τις διαφορές των δύο φύλων. Αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι να δούμε τα προβλήματα των προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου όπως είναι σήμερα και να πάρουμε τα κονδύλια για να τα πάμε εκεί που θα δαπανηθούν, εκεί που υπάρχουν καλά παραδείγματα από καλές πρακτικές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής. Σας ευχαριστώ και εγώ. Έχω την εντύπωση ότι τα προβλήματα δεν είναι τόσο ουσιαστικά έτσι όπως τα παρουσιάζετε εδώ και 39 χρόνια παρακολουθώ την περίπτωση των γυναικών που εργάζονται στον τομέα αυτό και έχω δει μεγάλες διαφορές. Πολλές περιπτώσεις υπάρχουν ε, γυναίκες που διαχειρίζονται, που ηγούνται σημαντικές, σημαντικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή είναι υπεύθυνε για τις πωλήσει. αγρονόμοι. Είναι μια νέα δραστηριότητα επαγγελματική. Αν θέλετε σημαντικά επαγγέλματα σήμερα εκπροσωπούνται από πολλές γυναίκες. Εγώ επί χρόνια ήμουν στην Εθνική Ομοσπονδία Γεωργών και όλο και περισσότερες γυναίκες συμμετείχαν όχι μόνο σαν μέλη της οργάνωσής μας αλλά και στο Συμβούλιο και σε πολλά καθαρά ανδρικά επαγγέλματα βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές γυναίκες. Οι γυναίκες σήμερα παίζουν όλο και λιγότερο χειρονακτικό ρόλο. Ένας ρόλος που σήμερα έχει αναλυφθεί από τα μηχανήματα, από τον εξοπλισμό. Βλέπουμε ότι οι γυναίκες περνάνε από προγράμματα κατάρτισης, είναι πιο μορφωμένες και χάρη στην τεχνολογία μπορούν να ασχοληθούν με άλλου είδους γεωργικά επαγγέλματα. Όντως, ε, συχνά ένα αγόρι είναι αυτό που αναλαμβάνει την ε, γεωργική εκμετάλλευση. Ένα κανονικό αγόρι κανονικά χρειάζεται και μία γυναίκα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εάν ο γεωργός θέλει να παντρευτεί και να έχει μία οικογένεια, η σύζυγός του μπορεί να παραμείνει στην γεωργική εκμετάλλευση, να συνεργαστεί, να εργαστεί, να διακόψει ενδεχομένως ε, όταν θελήσει να αποκτήσει παιδιά. Έτσι ακριβώς έκανε η γυναίκα μου όταν με παντρεύτηκε. Σήμερα βεβαίως είναι σύζυγος ευρωβουλευτή και μπορεί άνετα να συνεχίσει την γεωργική της δραστηριότητα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πριν προσλάβουμε κάποιον σε μια επιχείρηση ή σε μια γεωργική εκμετάλλευση κοιτάμε το φύλλο του. Κοιτάμε πολλά άλλα προσόντα. Εγώ παραδείγματο χάρη είχα προσλάβει μια γυναίκα στην, στο αγρόκτημά μου και μετά από λίγο καιρό η, η οικογενειακή της κατάσταση, ο σύζυγός της αποφάσισε να μετακομίσει και ορίστε που βρεθήκαμε. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα πρέπει να εξεταστούν και θα πρέπει να δούμε αν τα επιδόματα στηρίζουν ή οδηγούν του γεωργού να κάνουν κάποιε επιλογέ που θα τι είχαν κάνει αλλιώ. Δηλαδή αν εγώ έχω περισσότερη επιδότηση, αν προσλάβω γυναίκε, ε, αυτό θα με οδηγήσει ίσω σε κάποιε επιλογέ. Από την άλλη μεριά, εάν δεν προσλάβω του πιο αρμόδιου και αυτό θα με οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα. Θα σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ήταν ο τελευταίο μα ομιλητή, κ. Σάκνιου. Το λόγο λοιπόν θα έχει η κυρία Γέκλε και μετά οι προσκεκλημένε μα. Όχι, πρώτα οι Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε, αν θέλετε, στις ερωτήσεις. Πιο πολλές ερωτήσεις ε, αφορούν εμένα, οπότε ας ξεκινήσω εγώ. Να τις διατρέξω με τη σειρά. να σχολιάσω απλώς την τελευταία δήλωση, την τελευταία παρέμβαση. Γιατί υπάρχουν πολλά επιχειρήματα για το γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά εμείς κατά βάση θέτουμε το ερώτημα σε εσά. Γιατί εσείς θέτετε το, το θέμα του φίλου στα, όταν υπάρχει, υπάρχουν προτάσεις κομισιών, έγγραφα κλπ. Το θέμα του δεύτερου πυλώνα της ε, ΚΑΠ είναι πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαφοροποίησης, αγροπεριβαλλοντικά θέματα κλπ. Και σε όλα αυτά θα πρέπει να εξετάζουμε την σημασία των θεμάτων που τέθηκαν. Και Στράμπελα μίλησε για το θέμα της, ε, το, της περιουσιακής κατάστασης ε, των γυναικών και των ανδρών κλπ. Και σίγουρα χρειάζεται καλύτερη κατανόηση των ε, συμφωνιών και τι γίνεται με αυτές όταν επέρχεται διαζύγιο. Το θέμα αυτό ε, το ρυθμίζουν διαφορετικά νομοθετικά τα διάφορα κράτη-μέλη, χαρακτηρίζονται από διαφορετικές ε, παραδόσεις κλπ. Για την Ουγγαρία και την κοινωνία κράτη-μέλη επίσης ήταν πολύ σωστό το επιχείρημα. Και οι δυο μας είμαστε ποιοτικοί ερευνητές, ποιοτικές ερευνήστρες, δηλαδή ερευνούμε την ποιότητα και όχι τόσο πολύ την ποσότητα, μιλούμε με τους ανθρώπους. Παρόλα αυτά χρειαζόμαστε και ποσοτικά στοιχεία έτσι ώστε να γίνουν οι συγκρίσεις να είναι βάσιμες. Σίγουρα όμως πρέπει να κατανοήσουμε τη διαφορά ανάμεσα στα καινούργια και τα παλιά κράτη-μέλη και τη θέση της γυναίκας αυτά, καθώς επίσης και τις διαφορές ανάμεσα στα καινούργια κράτη-μέλη. Το λέμε επίσης τα έγγραφα ότι Δεν έχουμε σαφή στοιχεία για το ποιο είναι ο ρόλος των γυναικών σε μεγάλες βιομηχανικές εκμεταλλεύσει. Γι' αυτό το ζήτημα χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα. Σίγουρα. Τώρα, γιατί επιζητούμε αύξηση των γυναικών στη γεωργία. Χρειαζόμαστε ισορροπία πράγματι, όπως απαντήθηκε ήδη. Παρ' όλα αυτά το θέμα εξακολουθεί να είναι επίμαχο. Για τις συντάξεις των γυναικών και τη θέση των γυναικών μετά τη σύνταξη. Η νέα οδηγία την οποία αναφέραμε θα αλλάξει το τοπίο σε δύο χρόνια. Το πώς δηλαδή οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση στη σύνταξή τους. Γιατί τη Βόρεια Ιρλανδία είναι ενδιαφέρον το γεγονό ότι το 6% της ε, γεωργική, του γεωργικού δυναμικού κάτω των 40 είναι γυναίκες. Αλλά 12% είναι γυναίκες στο καινούριο project των νέων αφήξεων. Είναι πολύ καλά τα ποιοτικά αλλά και τα ποσοτικά στοιχεία βλέπετε είναι πολύ ενδιαφέροντα. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει περισσότερη γραφειοκρατία ή περισσότερη ρύθμιση, αλλά αυτό σίγουρα δεν σημαίνει πως από, λόγω του φόβου της γραφειοκρατίας πρέπει να αγνοήσουμε κάποια προβλήματα. Ε, είναι πολύ σημαντική επίσης η αύξηση ε, των, του αριθμού των γυναικών σε επαγγέλματα όπως ε, γεωπόνη, και κλπ. Δεν χρειάζεται γη για να μπουν όμως αυτά τα επαγγέλματα. Επίσης δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για να αποδείξουμε ότι οι γυναίκες ε, δεν οδηγούν μηχανήματα και δεν χειρίζονται μηχανήματα γιατί δεν τις εμπιστεύονται κλπ. Πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά εκεί. Ε, η γυναίκα σας είπατε διοικεί ε, την εκμετάλλευση. Ελπίζω να έχει, να, να έχει και την διοκτησία της. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο λόγος στην Πετίνα. Δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Να σας κάνω μερικά γενικά σχόλια καταρχήν. Γιατί είναι σημαντική η ισότητα των φύλων σε αγροτικές περιοχές. Πρώτον γιατί είναι θέμα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί η ισότητα είναι σημαντική αυτή καθ' αυτή. Αλλά ιδιαίτερα για την αγροτική ανάπτυξη και την κοινή αγροτική πολιτική ας θυμόμαστε ότι δεν είναι προς όφελος μόνο των γυναικών. Είναι προς όφελος και των ανδρών και προς όφελος της εδαφικής συνοχής και προς όφελος της ε, ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τον πληθυσμό ...από απομακρυσμένων περιοχών αν η ζωή τους δεν είναι ευχάριστη. Αν δεν είναι ευχάριστη η ζωή τους θα τις εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Δεν μπορούμε να τους καρφώσουμε εκεί πέρα. Αυτό ισχύει και για, τους, για γυναίκες και για τους άντρες. Και πολύ συχνά οι, τα αγόρια, οι νέοι, ε, είναι πιο δεδεμένοι με τη γη και έχουν λιγότερες δυνατότητες να φύγουν. Και πολύ συχνά μένουν ενώ φεύγουν οι γυναίκες. Και δεν έχουν και πολλές ευκαιρίες ενδεχομένως να βρουν θέση εργασίας αλλού γιατί δεν έχουν επενδύσει στην εκπαίδευσή τους. Συνεπώς είναι προς και των ανδρών να μένουν οι γυναίκες αλλά σίγουρα γενικότερα είναι προς όφελος της εδαφικής συνοχής. Τώρα, ποιοτική έρευνα, σημαντική ποιοτική έρευνα, αλλά τα ποιοτικά στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας δεν έχουν ε, δεν είναι ε, ισοκατανεμημένα. Έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία για τις παλιές χώρες, πολύ λιγότερα για τις καινούριες χώρες και σίγουρα πολύ λίγα στοιχεία για τις απομονωμένες ή περιοχές. περιοχές. Και υπάρχει λόγος. Γιατί, για παράδειγμα, οι απομονωμένες περιοχές ε, είναι λόγος από μόνες τους. Είναι δύσκολο κανείς να πάει εκεί και να κάνει την έρευνα. Έχουμε πολλά πράγματα για τα οποία υπάρχουν κενά και χρειάζεται να γίνει περισσότερη έρευνα και στατιστική έρευνα, αλλά κυρίως το σημαντικό είναι να καλύψουμε γεωγραφικά όλες τις χώρες και όλες τις περιοχές τους. Δεν ενδιαφέρει πιο πολύ η μελέτη της α ή της β περίπτωσης, μόνο περιπτωσιολογική μελέτη. Τα, η συνάδελφος από την Βόρεια Ιρλανδία είπε ότι οι οργανώσει παίζουν πολύ ρόλο, οι οργανώσεις γυναικών εννοώ, γιατί είναι σημαντικές και για την ίδια την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται, αλλά και για να κάνουν πιο ε, ακουστή τη φωνή των γυναικών στην κυβέρνηση. Στις κάτω χώρες οι γυναικέ οργανώσεις ε, υπάρχουν, αλλά αγωνίζονται για την επιβίωσή τους απλώς. Γιατί, γιατί όλο και λιγότερες γυναίκες θέλουν να γίνουν μέλη τέτοιων γυναικών οργανώσεων στην Ήπεθρο. Δεύτερον, διότι έχουν μικρή περιορισμένη χρηματοδότηση. Κάθε φορά πρέπει όλο και περισσότερα να, να σοφίζονται όλο και περισσότερα project για να εξασφαλίζουν χρηματοδότηση και θα μπορούσαν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν όντως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε και ελπίζω να μπορέσετε να συνεχίσετε την έρευνα την οποία έχετε ξεκινήσει σε αυτές τις πολύ απομακρυσμένες περιοχές. Αλλά θα τελικά το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Γέγκλερ για να μας συνοψίσει. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί σας απευθύνω το λόγο σε εσάς κυρία Πρόεδρε, ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας κανονικά είναι Άντρας. Πιστεύω ότι αυτό που μπορούμε να πούμε Καταρχήν είναι ότι δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους γεωργούς, από τις οικογένειές τους, στατιστικά στοιχεία και να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια. Γιατί πάντα αυτό είναι κάτι το γραφειοκρατικό, το δύσκολο. Από την άλλη μεριά βεβαίως ε, πολλές ερωτήσεις είναι χρήσιμες για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ορισμένα φαινόμενα. Η συζήτηση τελικά επικεντρώθηκε στην γυναίκα σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Υπάρχουν όμως και όλα τα άλλα τα συναφή με την ζωή και την δραστηριότητα των γυναικών στην Ήπεθρο. Αυτά με ενδιαφέρουν. Εγώ εργάστηκα 30 χρόνια σε μια γεωργική εκμετάλλευση. Όλα είναι σχετικά διότι εγώ μπόρεσα να ζήσω, να συνεχίσω τη δραστηριότητά μου και να κάνω και παιδιά. Οι γυναίκες τελικά αναλαμβάνουν πολλά βάρη γιατί τολμάνε να αναλάβουν όλα αυτά τα βάρη. Ζητώ λοιπόν από όλους τους συναδέλφους να επικεντρώσουν τη συζήτηση από εδώ και πέρα και την εργασία μας στη γυναίκα στην Ήπεθρο. Και εμείς είμαστε παρόντες σε θέματα δεύτερου πυλώνα. Δεν είναι μόνο θέματα περιφερειακής επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν σαφώς να πούμε ότι από τη μία υπάρχει το κοινωνικό ταμείο και η Ήπεθρος έχει πολλά και διαφορετικά φαινόμενα που τη χαρακτηρίζουν. Εμάς λοιπόν σαν Επιτροπή Γεωργίας μας αφορά άμεσα το θέμα αυτό της υπαίθρου και όλα αυτά που αφορούν το δεύτερο πυλώνα. Γνωρίζω ότι σε πολλά κράτη-μέλη σε θέματα δεύτερου πυλώνα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα που δίνουν σε ευκαιρίες στις γυναίκε. Στην Ιταλία παραδείγματο χάρη ξέρω ότι οι γυναίκες μπορούν στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις να οργανώσουν την φροντίδα των παιδιών και τη χρηματοδότηση αυτής της υπηρεσίας. Στην δική μου περιοχή στην Βαδιμουντεμπέργη υπάρχουν παρόμοια προγράμματα, το ίδιο και στην Αυστρία. Αυτά πρέπει να τα υπογραμμίσουμε, να τα συζητήσουμε, να τα παρουσιάσουμε σαν παραδείγματα, γιατί όλα αυτά κάνουν την Ήπεθρο ελκυστική για τους νέους, για τις γυναίκες. Γιατί αν εξαφανιστούν οι γυναίκες από τις περιοχές αυτές, καταλαβαίνετε ότι από δημογραφικής απόψεως το αποτέλεσμα είναι άμεσο. Είναι λοιπόν η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και είμαι πεπισμένη γι' αυτό. Έχω ήδη πολλές ε, γυναίκες ε, που μου στέλνουν προτάσεις και ιδέες, γυναίκες που είναι μέλη οργανώσεων. Εγώ ήδη ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Γεωργών, τότε που ήμουν δραστήρια και πραγματικά θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το γενικότερο πλαίσιο και επαναλαμβάνω πρέπει να πολεμήσουμε για τον δεύτερο πυλώνα στον προϋπολογισμό των γεωργικών. Όχι εδώ σε αυτή την Επιτροπή, γενικότερα. Γιατί υπάρχουν πολλά συμφέροντα, πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να πολεμήσουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την επεξεργασία αυτού του κειμένου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και ελπίζω να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τον ίδιο εξαιρετικό τρόπο. Ευχαριστώ. Τώρα θα κηρύξουμε τη λήξη της συνεδρίασης και θα αρχίσουμε αύριο στις 10 και με τους συντονιστές της 9. Η κοινή θνητή θα έρθουμε στις 10. It was okay.